Καλημέρα σας συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε τις εργασίες μας. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς την ημερήσια διάταξη, την εγκρίνουμε και ως προς τα πρακτικά της 16ης, 17ης Μαρτίου, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορούμε να τα εγκρίνουμε. Εγκρίνουμε λοιπόν τα πρακτικά σας ανακοινώνω ότι θα μαγνητοσκοπηθούν ένα μέρος των σημερινών μας εργασιών και θα προβληθεί αυτό το φιλμ στους ε, επισκέπτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω να μην υπάρχουν αντιρρήσεις για την παρουσία του τηλεοπτικού δικτύου και του δικτύου μαγνητοσκόπησης. Στη συνέχεια έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων με τον Ρόμπερτ Κούπερ, Γενικό Διευθυντή Εξωτερικών Υποθέσεων του, Ευρωπαϊκού, του Συμβουλίου, με σε σχέση με το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 26ης Απριλίου. Σας καλωσορίζω, δόκτωρα Κούπερ. Ήδη έχετε παρευρεθεί στις εργασίες μας για να μας μιλήσετε για την κατάσταση στο Ιράν. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 26 Απριλίου, ε, και θα μας πείτε τι διαδραματίστηκε όπως σας ζήτησε η ύπατη εκπρόσωπος, η κυρία Άστον. Θα ήθελα να επενθυμίσω στους ε, συναδέλφους ότι ο κύριος Κούπερ ε, αντικαθιστά την κυρία Άστον μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας επαφών και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και ΑΦΕΤ. Πρόκειται για την παγιωμένη διαδικασία μας και εκπροσωπεί την ύπατη εκπρόσωπο, την κυρία Άστον, όπως σας είπα. Ο κύριος Κούπερ θα παρέμβει και δεν θα μακρηγορήσει για να γίνει συζήτηση και θα μας μιλήσει για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και όχι Γενικών Υποθέσεων. Άρα δεν θα ασχοληθούμε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που προβλέπεται στο επόμενο σημείο που είναι ένα θέμα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων μέσα στα πλαίσια της ε, Ισπανικής Προεδρίας. Σας υπενθυμίζω λοιπόν τα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο. Καταρχήν τα συμπεράσματα σε σχέση με την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, την ΚΕΠΑ, και τις στρατιωτικές μας τρέχουσες δραστηριότητες. Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Πακιστάν και Αφγανιστάν, εκλογές στο Σουδάν και προκλήσεις και η κατάσταση στο Κυργιστάν. Δόκτωρα Κούπερ, σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ μαζί μας και σας δίνω το λόγο. Έχετε 15 λεπτά περίπου. Σα Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως είπατε, η ύπατη εκπρόσωπος που ταξιδεύει αυτή τη στιγμή μου ζήτησε να την αντικαταστήσω σε αυτή τη συνεδρίαση και θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να θεωρήσετε αυτή μια, ως μια μεταβατική διευθέτηση. Θα δούμε τι θα γίνει όταν συσταθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων την ε, προηγούμενη εβδομάδα, της 26ης δηλαδή, ήταν ε, μια ε, περίπλοκη πολυσχηδής διαδικασία, πολύπλευρη θα μπορούσα να πω, ήταν μια ξεχωριστή ε, συνεδρίαση μέσα στα πλαίσια της κοινή συνεδρίασης με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Υπουργούς Άμυνας. Υπήρχαν πολλά ουσιαστικά σημεία στην ουέσια διάταξη, όπως προείπατε, μεταξύ των οποίων και το Αφγανιστάν και το Σουδάν, Μιανμάρ, Βιρμανία, η κρίση στο Κυργιστάν και έγινε μια συζήτηση και για την Σομαλία. Όταν συναντήθηκαν οι Υπουργοί Άμυνας, συζήτησαν ως προς τις ε, τρέχουσες στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και θεσμικά και διαρθρωτικά ζητήματα που είναι απότοκα της προετοιμασίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. καθώς και τη συμμετοχή των Υπουργών Άμυνας στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Υποθέσεων ασχολήθηκαν με την στρατηγική ε, εξωτερικών σχέσεων Θα αρχίσω με την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας για να τα δούμε τα θέματα εν λεπτομερία, ασχολήθηκαν με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα ως προς την επιχείρηση Αταλάντα στις ακτές της Σομαλίας, τόνισαν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις πηγές της κακοδαιμονίας της πειρατείας, καθώς και την προστασία του στόλου. Η ύπατη εκπρόσωπος τόνισε την πρόθεσή της να επισκεφθεί την περιοχή για να ε, εξετάσει τι συμβαίνει, πώς δηλαδή εκτιλήσεται η επιχείρηση και τι συνέχεια θα δοθεί. Επίσης, οι Υπουργοί ασχολήθηκαν με μία ε, ε, επιχείρηση κατάρτισης στη Σομαλία έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το θέμα από ξηράς και θαλάσσης μέσα στα πλαίσια του συνολικού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την υποστήριξη της Σομαλίας. Τέλος, έγινε μία ανταλλαγή απόψεων ως προς το Άλτεα, δηλαδή την αποστολή μας στη Βοσνία όπου το θέμα της τέταρτης γενεάς είναι ένα ζήτημα ύψης της σημασίας οι Υπουργοί καλωσόρισαν την πρόθεση της ΥΠΑ της εκπροσώπου να γίνεται ε, συνάντηση σε τακτά χρονικά διαστήματα των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων με τους Υπουργούς Άμυνας σε θέματα, ως προς θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους καθώς και ενημέρωση των Υπουργών ως προς την κατάσταση της, ευρωπαϊκής, της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας εξωτερικής δράσης που θα συζητηθεί αργότερα. Τόνισε λοιπόν το γεγονός ότι μια τέτοια οργάνωση θα επέτρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια συνολική συνεκτική πολιτική και να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσει τα επιμέρους προβλήματα εξωτερικών υποθέσεων. Ως προς την συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων με τους Υπουργούς Άμυνας, ασχολήθηκαν με θέματα της θαλάσσιας ασφάλειας και κλήθηκαν τα κράτη-μέλη από την ύπατη εκπρόσωπο να εξεύρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν αυτό το περίπλοκο θέμα. Επίσης, η ύπατη εκπρόσωπος ενημέρωσε τους Υπουργούς ως προς την γενικότερη συλλογιστική μας ως προς την ε, απάντηση σε κατάστασεις, ε, επίγουσας ανάγκης και αυτό μετά βεβαίως το σεισμό της ΑΕΤΙΣ και το πώς τα κράτη-μέλη αντιμετώπισαν αυτή την κρίση. Οι Υπουργοί Άμυνας συζήτησαν και το ρόλο τους στην διαχείριση κρίσεων και ως προς την χρήση μηχανισμών άμυνας σε παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει και τους Υπουργούς Ανάπτυξης όταν ε, συζητούν στο ζήτημα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Και θα δούνε πώς μπορούν να ανταποκριθούν σε καταστάσεις φυσικών καταστροφών. Η κοινή συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών και Υπουργών Άμυνας χωρίστηκε σε δύο μέρη στο ένα συνεδρίασε το Συμβούλιο κάθε αυτό, όπου ασχολήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, το οποίο συμφωνήθηκε έξι μήνες πριν και μίλησαν για την απαρχή του σταδίου εφαρμογής αυτού του προγράμματος. Ο ε, πρέσβης Σάτσκας ε, διορίστηκε στην Καμπούλ ως εκπρόσωπος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει μεταβεί εκεί και μετά έγινε μια άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου όπου ο Γενικός Γραμματέας ε, του ΝΑΤΟ, ο κύριος Ράσμουσεν, είχε προσκληθεί και μας μίλησε για τη δραστηριότητα του ΝΑΤΟ. Έγινε μια συζήτηση ευρέως φάσματος ως προς τις δυνατότητες στενότερης συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Εθνών. Ε, όλοι έχουν νεοδιοριστέντες εκπροσώπους στο Αφγανιστάν πλέον και υπάρχει ε, δέσμευση και θέληση συνεργασίας. Μετά από τη συνεδρίαση αυτή και την έξοδο του Γενικού Γραμματέα, οι Υπουργοί Εξωτερικών μίλησαν για το Σουδάν μετά τις εκλογές που μόλις διενεργήθηκαν, αλλά οι συζητήσεις είχαν μία ε, προοπτική, μάλλον μία προβολή προς το μέλλον, διότι οι εκλογές αφορούν την ε, συνολική ειρηνευτική διαδικασία στην οποία προσδίδει μεγάλη σημασία το Συμβούλιο. Για το Σουδάν υπάρχουν, ε, ελοχεύουν πολύ κίνδυνοι βεβαίως, αλλά υπάρχει δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δράση. Ως προς το Κυργιστάν, η ύπατη εκπρόσωπος μας μίλησε στην ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατάσταση κρίσης και, τα, και οι υπουργοί έφτασαν σε συμπεράσματα έτσι ώστε να επανέλθει η, κατάσταση ειρήνης, δημόσιας τάξης και δημοκρατικής κυβέρνησης. Έτσι ώστε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια διαλόγου με τις νέες αρχές του Κυργιστάν, έτσι ώστε να τύχουν δημοκρατικής νομιμότητας εν ευθέτω χρόνο. Το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα ως προς τη Βυρμανία, ε, Μιανμάρ, τονίζοντας μεταξύ άλλων τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εκλογικό νόμο και διαβλέποντας δυνατότητες επίσκεψης ή αποστο... μιας αποστολής σε αυτή τη χώρα αργότερα μέσα στο έτος. Στα σημεία Α ελήφθη μία ε, απόφαση να επεκταθούν οι κυρώσεις για ένα ακόμα χρόνο να επεκταθεί το καθεστώς ε, κυρώσεων. Στα διάφορα, οι Υπουργοί Εξωτερικών επανήλθαν στο ζήτημα της επιχείρησης Ατλάντα για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της ε, πειρατείας και έγιναν συζητήσεις για επικείμενες αποφάσεις της κυβέρνησης της Κένιας έτσι ώστε να λήξει η συμφωνία για τη μεταφορά πειρατών η ύπατη εκπρόσωπος τόνισε την επιθυμία της να εξευρεθεί μια πλέον βιώσιμη λύση επί του θέματος. Και γι' αυτό ακριβώς θα επισκεφθεί την περιοχή στο εγγύς μέλλον. Και όπως σας είπα, οι Υπουργοί Εξωτερικών είχαν ανταλλαγές απόψεων για ε, στρατηγικές πολιτικές καθώς και κατανομή πόρων μεταξύ ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασικών εταίρων. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι αυτά είναι τα βασικά σημεία που συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και όπως είπατε και νωρίτερα το Συμβούλιο ενέκρινε ε, εκτενή συμπεράσματα για τις επιχειρήσεις CACP ως προς την ε, κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνας. Ευχαριστούμε, δόκτωρα Κούπερ. Εσείς ε, θέσατε επιτάπητο πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που θέλουν να παρέμβουν. Πριν ε, σας δώσω το λόγο, θα ήθελα να σας πω ότι επειδή πολλοί ζήτησαν το λόγο, ο χρόνος είναι περιορισμένος. Έχετε 1,5 λεπτό στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και δίνω το λόγο στον κύριο Σαλαφράγκα. Ε, ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον κύριο Κούπερ. Δεν είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε και όπως μας υπενθύμησε η σημερινή του παρουσία έχει προσωρινό χαρακτήρα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω όμως ότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα στο διευρυμένο Προεδρείο μετά από αίτημα τη δική μου ομάδας και άλλων πολιτικών ομάδων. Ήταν όντω πολύ μεστό το Συμβούλιο αυτό, η ημερήσια διάταξή του, ό,τι αφορά τη Σομαλία και την επιχείρηση Αταλάντη. Είναι πολύ σημαντικέ συμφωνίε με τρίτες χώρε για τη δίωξη των πειρατών. Αυτό φαίνεται και από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Μήπως θα μπορούσατε να μας αναλύσετε πιο διεξοδικά την παρούσα κατάσταση και πώς θα βελτιωθεί αυτό το θέμα στις σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κρίσεων, κύριε Πρόεδρε, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου κάνουν λόγο για την πιθανότητα έναρξης διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες και μερικές μάλιστα ήδη συμμετέχουν μαζί μας προκειμένου να γίνει δυνατή η συμμετοχή αυτών των τρίτων χωρών και αναφέρεται συγκεκριμένα η δυνατότητα συμμετοχής της Κίνας. Θα μπορούσατε να μας αναπτύξετε και αυτό το θέμα. Οι Κινέζοι το ζήτησαν ή πρόκειται για πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, διαπίστωσα ότι και για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας έγινε μία το στρατιωτικό δυνατοτήτων και ικανοτήτων. Θα ήθελα να μας κάνετε μία εκτενέστερη αξιολόγηση σε ό,τι αφορά την παρέμβαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Σας ευχαριστούμε κύριε Σαλαφράγκα. Το λόγο κύριος Σβάμποντα. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για θέματα ασφάλειας και άμυνας είχαμε χτες στην Υποεπιτροπή Άμυνας εντατική συζήτηση. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά λοιπόν. Όμως έχω τρία συγκεκριμένα ερωτήματα. Καταρχάς για τη Βοσνία. Συμμετάσχατε Στι συζητήσει για τη Βοσνία στο παρελθόν. Τώρα αναπτύσσονται νέε συνομιλίε και είπαν και οι Αμερικανοί από τη Washington την προηγούμενη εβδομάδα ότι προσπαθούν απλώ να διατηρήσουν την επικαιρότητα του θέματο. Πώ βλέπετε σε αυτέ τι νέε συνομιλίε για το συνταγματικό και τα λοιπά θέματα στη Βοσνία. Δεύτερον, αναφερθήκατε στην Κυργυσία. Ακούστηκε από την Γερμανική Προεδρία η ιδέα της ανάπτυξης μιας κεντρο ε, μια στρατηγική για την Κεντρική Ασία δεν ε, αφορούν τα προβλήματα μόνο μία χώρα στη τελευταία ανάλυση, αλλά μια ολόκληρη περιοχή. Θα αναζωογονηθεί λοιπόν αυτή η προσπάθεια και θα καλύψει τις άλλες χώρες. Τέταρτον, βλέπω ότι δεν, ακούγεται λόγος, δεν έχει γίνει λόγος για το Ιράν στη συζητήση των υπουργών των εξωτερικών. Ενώ από την επίσκεψη στη Washington είχαμε ακούσει ότι υπήρχε μια πρόταση για κυρώσεις σε επίπεδο Κογκρέσου παρά τις διμερείς προσπάθειες της κυβέρνησης και στη συνέχεια όποια χώρα δεν ακολουθούσε τις κυρώσεις που είχαν προτείνει οι Αμερικανοί, το Αμερικανικό Κογκρέσο, θα εφίσατο με την σειρά της κυρώσεις. Για μονομερή ανάληψη δράσης κτλ. Ε, πράγμα το οποίο φυσικά θα έπλητε και τις ευρωπαϊκές χώρες. Γνωρίζουν αυτά τα ζητήματα οι υπηρεσίες σας, οι υπηρεσίες των εξωτερικών υποθέσεων. Ε, είναι ενήμεροι οι υπουργοί των εξωτερικών, ότι υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ε, επιβληθούν κυρώσεις για μονομερή ανάληψη δράσης ε, στα ευρωπαϊκά κράτη. Ο κύριος Βότσον, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να σημειώσω ότι θα ήταν σκόπιμο πιο τακτικά να συνεδριάζουν οι Υπουργοί των Εξωτερικών και βέβαια με την ύπατη εκπρόσωπο. Και αν μου επιτρέπει ο κύριο Σκούπερ να διατυπώσω πιο συγκεκριμένε ερωτήσει, η μία φορά το Αφγανιστάν, μιλήσατε για την ΑΦΠΑΚ. Η ΠΑΚΑΦ, ε, δεδομένη και τη ιδιαίτερα εκρηκτική κατάσταση στο Αφγανιστάν, πρέπει να, στο Πακιστάν, πρέπει να το δώσουμε και αυτούν την προτεραιότητα, όχι μόνο στο Αφγανιστάν, τουλάχιστον αυτό πιστεύει η ομάδα μου. Και για τα σχέδια των Υπουργών Άμυνας, να συγχωνεύσουν τουλάχιστον να στήσουν μια καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν και το, της επίσκεψης της ε, ρωτάτης Εκπροσώπου στην Ινδία στις επόμενες εβδομάδες είναι κάτι το οποίο θα συζητήσει, θα θέσει στους ε, ομολόγους της επίπεδο ΝΑΤΟ και επίσης τις ε, λεγόμενες ε, έξω δικαιικές εκτελέσεις, οποίες είναι εμπλεγμένοι οι Αμερικανοί με την, προσπάθεια, με την προτίμηση όπως γνωρίζετε που έχουν μερικές φορές ε, να εκτελούν ε, φερρυπίν φερόμενα μέλη της Αλκάιντα προκειμένου να χρειαστεί να τα προσαγάγουν σε δίκη. Έχει αναλυφθεί κάποια δράση στην υπόθεση αυτή, έχει κανείς να λάβει πρωτοβουλία και επίσης είδαμε και κάποιες νόμιμες στο ΣΥΠΗΝ ε, εκτελέσεις στην Ταϊβάν που ξανάρχισε να εκτελεί πολίτες, όχι βέβαια στο βαθμό που τους εκτελεί η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, αλλά εκτελεί ε, θανατικές ποινές και θα ήθελα προκειμένου να υποστηρίξω τις δηλώσεις της ΥΠΑ εκπροσώπου ε, που προσβάλλουν αυτή, την, που επιτίθεται κατά αυτής της υπόθεσης. Κύριε Λοντσέκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να, εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έλευση του κυρίου Κούπερ για να μας αναλύσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της προηγούμενης εβδομάδας. Ευελπιστώ όμως ότι στο μέλλον καλό θα ήταν να έχουμε είτε εσάς την κυρία Άστον αμέσως μετά τέτοιες ε, συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Πάντως χαίρομαι ιδιαίτερα που ήρθατε έστω και σήμερα. Σε ό,τι αφορά αυτά που ρώτησε ο κύριο Βόμποντα για τη στρατηγική για την Κεντρική Ασία, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί από το Συμβούλιο. Και σε ό,τι αφορά την ε, αποστολή Γιούλεξ. είμαι συγκέντρια για το Κωσυφοπέδιο και άρτη αφιχθήσα από αποστολή εκεί. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία που είχα στο Κωσυφοπέδιο όταν άρχισε η Γιούλεξ κάποιε έρευνε σε υψηλό επίπεδο στο Υπουργείο Μεταφορών και ορισμένες, ορισμένων σκανδάλων διαφθοράς και δωροδοκίας. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ανέφεραν την ανάγκη της συμμετοχής της ε, Γιούλεξ στην έρευνα και δίωξη σημαντικών υποθέσεων τέτοιων περιπτώσεων διαφθοράς. Χαίρομαι που άρχισε μια τέτοια διαδικασία και μάλιστα σε υψηλά κλιμάκια, γιατί υπήρχαν κατηγορίες ε, κατά υψηλό βαθμό αξιωματούχων για εμπλοκή τους σε σκάνδαλα διαφθοράς. Ίσως όμως ε, η Γιούλεξ αντιμετωπίσει προβλήματα με κάποιες άλλες α, ε, ίσως με τις Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί ίσως για τι τις Πολιτείε υπήρχε υπήρχε άλλη διέξοδος από ότι αυτή που κατέληξαν ο κ. Σάτσι και η Γιούλεξ. Τι γνώμη έχετε για την ε, παράταση της εντολής της Γιούλεξ. Ποια είναι η θέση του Συμβούλου αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πρόταση για υποστήριξη και ενίσχυση της πρόοδου της Γιούλεξ για να καταπολεμήσει τους καρχαρίες, όπως λέμε, της διαφθοράς στο κοσυφοπαίδιο. Και η τελευταία παρέμβαση από την πρώτη ομάδα ερωτήσεων, η κυρία Λέζινγκ. Παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο αγόρευσης που είναι 1,5 λεπτό, γιατί περιμένουν και άλλοι συνάδελφοι να μιλήσουν. Οι άλλοι μίλησαν από δύο λεπτά, αν μου δίνατε και εμένα. Καλά θα ήταν, εν πάση περιπτώσει, περιοριστώ σε αυτά. Κύριε Κούπερ, στο 88 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου διαβάζω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατυπώνει προτάσεις για εντατικοποίηση των ε, συνεργασιών με τον ΝΑΤΟ. Αλλά κάτι συγκεκριμένο δεν είδα πουθενά. Τι περιλαμβάνουν αυτές οι προτάσεις. Είναι δημόσιες. Μπορεί κανείς να τις ε, συμβουλευτεί και πότε θα ενημερωθούν επισήμως οι βουλευτές. Στο 16 επίσης των συμπειρασμάτων αναφέρεται η πρόσφατα ε, εγκαινιστή σα συνεργασία για το Αφγανιστάν με το ΝΑΤΟ. Με πολύ εγκομιαστικά λόγια. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιο βαθμό εκτείνεται αυτή η συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Και επίσης το 6 γίνεται λόγος για το κοσφοπέδιο και την ε, απόρριψη από τις σερβικές οικογένειες που ζουν εκεί, αλλά και τη σερβική κυβέρνηση των προτάσεων. Ε, αυτό το έχουν συζητήσει όντως με, τους, με τους Σέρβους ή όχι. Υποστήριξη για την προσέγγιση της αποστολής. Ευχαριστώ. Το λόγο για ο Δόκτωρ Κούπερ για να απαντήσει τις πρώτες πέντε παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ καταρχήν στις ερωτήσεις του κυρίου Σαλαφράγκα για τη Σομαλία και τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Φυσικά υπάρχουν δύο κατηγορίες τρίτων χωρών και ανάμιξη τρίτων χωρών. Υπάρχουν χώρες που συνεργάζονται στις επιχειρήσεις μας και υπάρχουν και οι ρυθμίσεις που έχουμε επεξηράσει με κάποιες χώρες για τη δίωξη των πιλωτών. Και η δεύτερη κατηγορία μας απασχόλησε ιδιαίτερα. Και στο πλαίσιο αυτό ε, είχαμε επαφές με διάφορες χώρες. Για παράδειγμα έχουμε ρυθμίσεις με την Κένια, με τις Αιχέλες, το Μαυρίκιο, την ε, Νότια Αφρική, την Ταζανία, την Ουγκάντα. Είχαμε επαφές με όλες αυτές τις χώρες, ε, διερευνώντας τη δυνατότητα σύναψη συμφωνιών για ένα ευρύτερο καταμερισμό ευθυνών στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συνεργασία στις ε, επιχειρήσεις του ναυτικού, ο κύριος Σαλαφράνκα αναφέρθηκε στην Κίνα. Υπάρχει συνεχή συνεργασία με την Κίνα. Γιατί υπάρχει και ένα κινέζικο σκάφος εκεί στην περιοχή που έχει τακτικές επαφές με το Γενικό Επιτελείο των Επιχειρήσεων. Οπότε υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και αυτό ισχύει όχι μόνο για την Κίνα αλλά και για την Ιαπωνία. Και εκεί οι πληροφορίες από αεροσκάφη της ε, Ιαπωνίας είναι πολύ σημαντικά για την περιοχή και είναι σημαντικές αυτές οι πληροφορίες για όλες τις χώρες που έχουν πλοία στην περιοχή. Για μας είναι η πρώτη φορά που έχουμε άμεσες ε, στρατιωτικές επαφές με την Κίνα και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, χρήσιμο και επικοδομητικό. Και δείχνει πόσο η αναγνώριση της μάστιγας της ε, πειρατείας απασχολεί τους πάντες. Γιατί όντως ε, προβληματίζει όλες τις χώρες. Σε ό,τι αφορά κυρία Σβόμποντα τη Βοσνία, αναφέρθηκε η επιχείρηση Αλτέα στα συμπεράσματα, αλλά δεν ε, περιλήφθηκε η Βοσνία στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Ειλικρινά σας λέω, οι προπτικές ε, επίτευξης προόδου σε μια δυστυχώ προεκλογική κατάσταση στη Βοσνία δεν είναι και πολύ λαμπρέ. Η πιο επικοδομητική προσέγγιση ίσως θα ήταν διακριτικές επαφές με τους ενδιαφερόμενους για να δούμε τι μπορεί να γίνει μετά τις εκλογές. Αυτά ως προς το που στέκει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Για την Κυργυζία, Κυργιστάν και την στρατηγική της Κεντρικής Ασίας ε, ισχύει αυτή η στρατηγική. Τουλάχιστον υπάρχει εστίαση στο, στην Κεντρική Ασία και η Πία έχει παρουσία στην περιοχή και μόλις εκδηλώθηκαν τα συμβάντα στο Κυργιστάν, στην Κυργιζία υπήρξε άμεση μετάβαση. Θα συνεχιστεί λοιπόν η πρόσοχή μας προς την περιοχή αυτή. Και σίγουρα η εξελίξη σε μία περιοχή έχουν άμεσο αντίκτυπο και στις γειτονικές, στις γειτονικές χώρες. Ο κύριος Βόμποντα αναφέρθηκε στην παράληψη του Ιράν από την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Υπουργών το Ιράν θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου της επόμενης εβδομάδας, γιατί ήταν παραφορτωμένη η ημερήσια διάταξη της προηγούμενης εβδομάδας, γι' αυτό προτιμήσαμε να μεταθέσουμε το Ιράν στο πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας. Δεν συζητήθηκε λοιπόν το Ιράν, αλλά η ύπατη εκπρόσωπος έστειλε επιστολή στον ε, στην Αμερικανίδα Υπουργό Εξωτερικών σε ότι αφορά το ψήφισμα του Κογκρέσου και την ανάγκη ενίσχυση συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, καθώς και την διαμαρτυρία μας, την αντίρρησή μας ό,τι αφορά την ανάληψη μονόπλευρης δράσης, μονομέρους δράσης. Σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις του κ. Βότσαν για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, εκεί η συζήτηση για το Πακιστάν δεν επισήλθε στην ουσία. Γιατί ενέσκυψε ο σεισμός και έτσι δεν υπήρξε η αναμενόμενη συνάντηση. Νομίζω ότι για το Αφγανιστάν θα πρέπει να οργανώσουμε ένα ορθολογικό καταμερισμό του φόρτου εργασίας. Και η παρουσίαση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ δείχνει την σπουδαιότητα που προσδίδουμε στη συνεργασία αυτή με τον ΝΑΤΟ και υπάρχουν τακτικές επαφές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή ε, έχει αναπτύξει εκεί πολύ σημαντική ειρηνευτική αποστολή, αλλά αυτά που κάνει το ΝΑΤΟ και αυτά που κάνει η UPOL στην πράξη συνδυάζονται θαυμάσια το ΝΑΤΟ ασχολείται περισσότερο με την ε, αστυνομία και η UPOL ε, ασχολείται με θέματα οργανωτικά σε επίπεδο επιτελείου, θέματα ερευνητικά, θέματα κατάρτισης αστυνομίας, γιατί η αστυνομία είναι σχεδόν έχει στρατητικό χαρακτήρα. Οπότε χρειαζόμαστε και μια αστυνομία που πραγματικά θα καταπολεμά το έγκλημα. Γιατί στο Αφγανιστάν υπάρχει πολύ εξίσου σημαντικό κίνδυνο να απεχθεί κανεί από εγκληματίε από ότι να χάσει τη ζωή του από μια βομβιστική ενέργεια των τρομοκρατών. Οπότε θα πρέπει να αναπτυχθεί και αυτή η δυνατότητα τη αστυνομία πραγματικά να καταπολεμά το έγκλημα. Σε ό,τι αφορά την Ινδία. Ο ρόλος της Ινδίας στο Αφγανιστάν ήταν ανέκαθεν σημαντικός. Και επίσης είναι σημαντικό να αποφευθούν παρεξηγήσεις ως προς τον ρόλο της Ινδίας στο Πακιστάν σε σχέση με άλλες δυνάμεις της περιοχής στο Πακιστάν. Το θέμα των εξώδικων εκτελέσεων ή δολοφονιών θα ήθελα να το παρακάμψω, γιατί δεν συζητήθηκε από τους υπουργού. Ίσως ε, συζητάτε περισσότερο στο ΝΑΤΟ παρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, θα έπρεπε να το είχα πει ίσως στην αρχή. Είπα ότι λυπούμε που ήρθε αυτή τη βδομάδα και όχι αμέσως μετά το Συμβούλιο, την προηγούμενη βδομάδα. Αλλά αμέσως μετά το Συμβούλιο η είπατε εκπρόσωπο έφυγε για την Άπο Ανατολή και τη συνόδευσα σε αυτή την επίσκεψη. Γι' αυτό δεν μπόρεσα να έρθω μαζί σας, στην να έρθω στην συνεδρίαση την προηγούμενη εβδομάδα και ζήτησα συγγνώμη γι' αυτό. Ως προς τις ερωτήσεις της κυρίας Λούνατσεκ. Το θέμα της Γιούλεξ. Συμφωνώ μαζί σας κυρία Λούνατσεκ ότι είναι θετικό που η Γιούλεξ ήδη έχει αναλάβει δράση σε θέματα πάταξης της διαφθοράς. Και σίγουρα το πιο συνετό θα ήταν να πω ότι συμμερίζομαι τη γνώμη της ότι το θέμα αυτό είναι πολύ λεπτό. Μια και μερικές φορές υπάρχουν διαπλοκές εγκλήματος και πολιτικού κόσμου. Σε ό,τι αφορά τη Γιούλεξ, υπάρχουν φυσικά δικαστές και εισαγγελείς που αυτοί να βαλαβάνουν τις απο, αποφάσεις με βάση τα τεκμήρια που συλλέγουν, τις αποδείξεις που συγκεντρώνουν, ανεξάρτητα ε, ενεργούν και διώκουν εγκλήματα όταν πιστεύουν ότι υπάρχουν ε, βάσιμα τεκμήρια που στοιχειοθετούν την διάπραξη ενός εγκλήματος και το τεκμηριώνουν. Από ό,τι Βλέπω, έχετε στην ημερήσια σας διάταξη συζήτηση για το πεδίο αργότερα και επευκαιρία της ε, αξιόλογης έκθεσης σα, κυρία Λούνατσεκ. Σε ό,τι αφορά τι ερωτήσει της κυρία Λόζινγκ για τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ulex και της Ιούπολ, αυτά είναι σε θέματα ειρηνευτικά κυρίω και συμφωνήσαμε με τον κύριο Ράσμουσεν ότι υπάρχει καλό συντέργεσμα των ε, δραστηριοτήτων της UPOL με τις ε, δραστηριότητες του ΝΑΤΟ. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη προστασία και να επεκτείνουμε ίσως το έργο της UPOL και να ε, επεκτείνουμε την ε, τάξη και σε αστικά κέντρα πέρα της Καμπούλ, γιατί μέχρι στιγμής είχαμε επικεντρωθεί στην Καμπούλ. Έχω την αίσθηση ότι οι γενικές εξελίξεις είναι μάλλον θετικές και οι περισσότεροι κάτοικοι του Βορρά έχουν διαπιστώσει ότι δεν ισχύει και πολύ ε, το κράτος δικαίου και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και φυσικά ε, οι άνθρωποι χρειάζονται κάποια νομική ασφάλεια σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία για παράδειγμα, τι γίνεται σε περίπτωση ενός ατυχήματος ε, τροχαίου. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία και Γενικώ ο τοπικό πληθυσμό καλωσόρισε την επέκταση των δραστηριοτήτων τη Γιούλεξ και προ το βορρά. Ευχαριστούμε, δόκτωρα Κούπερ. Περνάμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Σλέφλιν. Νομίζω, Νομίζω ότι εννοείται εμένα μάλλον. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος, δεν είμαι πολύ καλός στην προφορά ξέρω ονομάτων. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, κατάλαβα αρκεί αυτό. Ευχαριστώ τον Δόκτωρα Κούπερ για την παρουσία του εδώ. Αναφερθήκατε στο ρόλο της Κίνας, αλλά εν γέννη. Πώς βλέπετε το ρόλο της Κίνας σε σχέση με τις ε, δραστηριότητες, ε, τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη βλέπετε να υποστηρίζει αυτές τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες, να, να αντιστέκεται, να αντιδρά ή να είναι αδιάφορη. Σύντομη ερώτηση, λέει ο Ευχαριστώ. Και θα δώσω το λόγο τώρα στον συνάδελφο Βάγγελ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Στην Επιτροπή Ανάπτυξης και χάρη στην όθηση που μας έδωσε ένας από τους συναδέλφους με τις πρωτοβουλίες του. Συζητήσαμε τα ε, θέματα που μοιάζουν με αυτά που μας απασχολούν σήμερα εδώ και πρέπει να πω ότι καταλήξαμε πως θα πρέπει στα συμπεράσματα του Συμβουλίου να αναζητούμε περισσότερο το περιεχόμενο και όχι τις τεχνικές πληροφορίες. Και έτσι, κύριε Κούπερ, σε αυτήν την πρώτη ε, συζήτηση αυτό το πρώτο γύρο ερωτήσεων. Μας δώσατε πολύ ουσιαστικές ερωτήσεις και γι' αυτό σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Ιδιαίτερα μα διαφωτίσατε δε για τα θέματα της βοσνίας Ερζεγοβίνη αλλά και άλλα. Και πάνω απ' όλα είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε προς τα πού πλέει το σκάφος. Έχουμε μια εικόνα του ε, πού πηγαίνουμε και ποια θα είναι η παρουσία η δική μα εκεί. Επίσης θα πρέπει να επανεξετάσουμε άλλε αποστολές στη Γουινέα Βισάου. Έχουμε μία αποστολή η οποία είναι περίτη, δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξη, πρέπει να καταργηθεί. Στο κοσμοπέδιο χρειάζεται μια νέα πολιτική ανάλυση της κατάστασης. Υπάρχουν άλλοι τομεί στου οποίου χρειαζόμαστε περισσότερο περιεχόμενο, περισσότερη ουσία. Ευχαριστώ. Λόχμπιλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Κούπερ για την εκθέση σας. Έχω δύο πολύ στομές ερωτήσεις. Πρώτον, ε, την ε, διεθνή διάσκεψη για την αναθεώρηση του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου που θα ξεκινήσει 31 Μαΐου από την Επιτροπή για τα Ανθρωπινά Δικαιώματα έχουμε ενημερωθεί για την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων αλλά έχουμε επίσης ενημερωθεί ότι δεν επιτυγχάνεται συμφωνία σε διάφορα θέματα σημαντικά Όπω σε παραδείγματι το ζήτημα ενό επιθετικού πολέμου. πώ θα το χειριστεί αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα είναι αυτή η διάσκεψη λοιπόν. Θα είναι απλώ μια διάσκεψη καταγραφή τη κατάσταση, δεν θα είναι και μια πολιτική κατάσταση, θα χειριστεί τα θέματα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει υποστηρίξει ολόκληρη το ε, διεθνέ Δικαστήριο Ποινικού Δικαίου να ε, ε, είναι παρούσα με σαφείς θέσεις και για τη δεύτερη ερώτηση το Ιράν, που είπατε ότι θα σας απασχολήσει την προσεχή εβδομάδα, θα ήθελα να μάθω ποιος πρόκειται να συμμετάσχει στην διαπραγματευτική ομάδα για τα πυρηνικά του Ιράν. Όπως ε, το έκανε ο κύριος Σολάνα στο παρελθόν, σκοπεύει μήπως και η Λέδη Άστον να αναλάβει την πρωτοβουλία και την ηγεσία, την ηγετική, τον ρόλο σε αυτήν την ομάδα. Μπρέντα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ, κύριε Κούπερ. Μια ερώτηση μόνο, που αφορά την Βυρμανία, Μιανμάρ. Υπάρχει στα συμπεράσματα του Συμβουλίου η πρόθεση της αποστολής μιας ε, ε ομάδας. Τι θα γίνει λοιπόν εκεί, θα γίνουν οι εκλογές ή θα αναβληθούν επειδή ο εκλογικός νόμος δεν αρκεί για την εξαγωγή απρόσκοπτων και δίκαιων εκλογών ή θα παραταθεί μια προεκλογική περίοδος για να καταλήξουμε στις εκλογές ενδεχομένως πάλι μέσα στο 2010 αλλά πιο αργά. Είναι πολύ σημαντικό να γίνουν οι εκλογές εκείνη. Ας δώσουμε χρόνο στον συνάδελφο Σάκε. Συνάδελφο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κούπερ και εγώ με τη σειρά μου και εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω για το Ιράν. Καθίσταται σαφές ότι το ζήτημα αυτό ε, είναι ένα έντονο ζήτημα και την προηγούμενη ε, εβδομάδα που παρευρέθηκα στην Ουάσιγκτον ε, μίλησα με μέλη της Γερουσίας. Πιστεύω ότι είναι περίεργη ιδέα να αναβάλουμε το ζήτημα στην για την επόμενη εβδομάδα, διότι πολλά διαδραματίστηκαν αυτή την εβδομάδα. στο θέμα των πυρηνικών, ο Αχμαντινετζάντ ε, έθεσε ορισμένα ζητήματα. Αξιωματούχοι του Ιράν ε, μετέβησαν στις ΗΠΑ. Επίσης, στο, στα Ηνωμένα Έθνη, στο Συμβούλιο Γυναικών, υπήρξαν δυσκολίες και ίσως με αυτή την ευκαιρία θα μπορούσαμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή θέση σε αυτά τα θέματα ύψης της σημασίας. Όταν παρευρέθηκα στη Γερουσία την προηγούμενη εβδομάδα, και οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκράτες ε, είναι υπέρ των μονομερών κυρώσεων και ε, στυλιτεύουν την σιωπή της Ευρώπης. Δεν πρέπει να δώσουμε τροφή σε αυτή τη ρητορική. Τον είπα και πιστεύω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε με μία φωνή, διότι το θέμα των πυρηνικών και του Ιράν είναι μείζονο σημασίας. Θα ήθελα να σας προτρέψω λοιπόν να συνεργαστείτε με το Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα ζωτικής σημασίας και θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο η Τουρκία θα μπορούσε να διαδραματίσει κάποιο ρόλο και πώς θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε την Τουρκία έναντι του Ιράν επί του θέματος αυτού. Ο δόκτωρ Κούπερ έχει το λόγο, θα ήθελα να περιοριστείτε ως προς το χρόνο, έτσι ώστε να έχουμε και τον τελευταίο γύρο ερωτήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος όπως ήταν και ο, η κυρία Σέπλιν. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αν και δεν σχετίζονται όλες με τις παρεμβάσεις του Συμβουλίου. Στον κύριο Σέπλιν θα ήθελα να πω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με το, με το Συμβούλιο, αλλά επειδή μετέβην στην Κίνα με την Λέδη Άστον την προηγούμενη εβδομάδα, μπορώ να σας πω ότι υπάρχει πολύ θετική στάση της Κίνας για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που μας απασχολεί. Ε, θετική στάση, αλλά κάπως απόμακρη. Γι' αυτό υπάρχει ε, κοινό πεδίο δράσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις, ε, την έμπρακτη πτυχή πολλών θεμάτων. Και βεβαίως ε, αυτό αφορά και το Αφγανιστάν που είναι μια ε, γείτον χώρα. Συζητήσαμε το θέμα με την Κίνα καθώς και το θέμα της ε, Σομαλίας και του Σουδάν. Γιατί ξέρετε ότι η Κίνα έχει επαφές με αυτές τις χώρες και έχει νόημα να αρχίσουμε ένα διάλογο. Ως προς το ερώτημα του κυρίου Βάγκελ, είμαι κάπως επιφυλακτικός. Δεν θα ήθελα να προβώ σε μία ανάλυση της πολιτικής κατάστασης στη Βοσνία, που είναι περίπλοκη και καθόλου ικανοποιητική ακόμα. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία ενός θετικού ε, αντικτύπου της απόφασης του Κοινοβουλίου στη Σερβία που πρόθεσε ο πρόεδρος Τάντιτς ε, μιλώντας για τη δέσμευση της Βοσνίας έναντι, έναντι θεμάτων εδαφικής κυριαρχίας. Αλλά αυτά τα θέματα προέρχονται εκτός Βοσνίας και όχι εντός. Θα ήθελα υπό άλλες συνθήκες να το συζητήσουμε λεπτομερέστερα. Ως προς τη Γουινέα Μπισάου, θα ήθελα να πω ότι αναθεωρούμε την ε, θέση μας ως προς την αποστολή εκεί. Υπάρχει ένας ε, αριθμός κινδύνων στη Δυτική Αφρική ως προς τη διακίνηση ναρκωτικών και θα θέλαμε να βρούμε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης παρόμοιων χαοδών καταστάσεων. Για την κυρία Λόχμπιλερ, ως προς το ερώτημα της, το θέμα του ICC δεν συζητήθηκε στο Συμβούλιο. E Από όσο γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει το ICC αλλά και εγώ δεν γνωρίζω τα τελευταία δεδομένα της διάσκεψης. Um, uh, Αυτά ως προς το διεθνές ποινικό. Ε, υπήρξαν και δύο ερωτήματα για το Ιράν. Ως προς τον χρονισμό, πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία στο Ιράν. Συζητείται μερικές φορές στο Συμβούλιο και πολύ συχνά uh, um, στο PSE και φαίνεται ότι υπάρχει μια συνεχής ροή γεγονότων και συμβάντων και θα θέλαμε μια πιο διεξοδική συζήτηση επί του θέματος. Η Κάθριν Άστον στη Νέα Υόρκη ε, ασχολήθηκε με το θέμα της διάδοσης των πυρηνικών όπλων στο, ως προς το μηχανισμό NPT και το έχει συζητήσει και στην Κίνα. Σε σχέση με το ε, ερώτημα της κυρίας Σάρκα, έχει συνομιλήσει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Πρόκειται λοιπόν για μια συνεχή διαδικασία της ε, πολιτικής μας, διότι προσδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτό το σκέλος. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή οι διαπραγματεύσεις με τους ε, Ιρανούς θα αναβιώσουν. Και οι κυρώσεις υπάρχουν για να υπενθυμίσουμε στους Ιρανούς ότι θέλουμε να επιληθεί το θέμα αυτό μέσα από διαπραγματεύσεις και συμφωνία. Και οι κυρώσεις υπάρχουν για να επισύρουμε την προσοχή του Ιράν στο γεγονός ότι αν δεν διευθετηθεί το θέμα μέσω συμφωνίας, θα πρέπει να εξεύρουμε άλλους τρόπους για να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η επιθυμία μας λοιπόν είναι να επανέλθουμε στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων με τους Ιρανούς το ταχύτερο δυνατόν, όποτε εκείνοι είναι έτοιμοι να συζητήσουν το, την ουσία του θέματος. Και κατά τις προσδοκίες μου, αν επισυμβεί κάτι τέτοιο, η Κάθριν Άστον θα αναλάβει το ρόλο του Χαβιέ Σολάνα στο παρελθόν. Θα έχουμε 3 συν 3, 5 συν 1. Κατά πόσο θα επηρεαστεί αυτός ο μηχανισμός από τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, δεν το ξέρω. Μιλάμε για 3 συν 3 ή 5 συν 1. Ίσως θα πρέπει να μιλάμε για 3 συν 3 συν 1, διότι υπάρχουν 6 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Πρέντα υπέβαλε ένα ερώτημα για την διερευνητική αποστολή στη Βυρμανία. Θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχουν μεγάλες ελπίδες να ανατρέψουμε τον εκλογικό νόμο. Η διερευνητική αποστολή ήρθε σε επαφή με τα πολιτικά κόμματα και όχι μόνο με κυβερνητικούς εκπροσώπους. Προσπαθούμε να ε, αυξήσουμε τις ε, επαφές μας, διότι εδώ και πολύ καιρό δεν είχε μεταβεί καμία αποστολή στη Βυρμανία και θέλουμε να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς της Βυρμανίας που αποζητούν ένα δημοκρατικό μέλλον και συμφιλίωση. Νομίζω ότι απάντησα εν μέρη το ερώτημα της κυρίας Σάρκα. Θα ήθελα να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι στο Ιράν εδώ, πέντε, εδώ και 5-6 χρόνια και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλές περιστάσεις ενίσχυσε τις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών. Δυστυχώς αυτά τα νέα δεν έφτασαν μέχρι την Ουάσιγκτον, τουλάχιστον όχι μέχρι το Κογκρέσο. Και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε η θέση μας, που είναι παρόμοια με της κυβέρνηση των ΗΠΑ, να γίνει απόλυτα κατανοητή. Ως προς την Τουρκία, η τουρκική κυβέρνηση, ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός είναι γείτονες του Ιράν, γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν. Θεωρώ ότι οι συμβουλές τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και με αυτά τα δεδομένα η Κάθριν Άστον είχε μακρές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Άρα παραμένουμε πολύ κοντά ε, στη θέση της Τουρκίας, αν και δεν συμφωνούμε απόλυτα με τον πολιτικό λόγο της Τουρκίας. Ευχαριστώ. Η τελευταία, τώρα τελευταίος γύρος των παρεμβάσεων. Η συνάδελφος Γκόμες έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Κούπερ. Έμεινα άναυδη με τη δήλωση του Συμβουλίου για τις εκλογές στο Σουδάν. Δεν ανταποκρίνεται καθόλου ούτε με την κοινοβουλευτική μέσα αποστολή και τα συμπεράσματά της, ούτε με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δήλωνε ότι σε καμία περίπτωση οι εκλογές στο Σουδάν δεν ε, πληρούσαν τις διεθνείς προδιαγραφές για ανώθευτες εκλογές. Παρά είναι χαλαρή και ήπια η δήλωση του Συμβουλίου γι' αυτό. Και πολύ φοβάμαι ότι πολύ σωστά όταν ο επικεφαλής παρατηρητής αποφάσισε να αποσύρει τους δικούς μας παρατηρητές από τον Ταρφούρ, τότε συντάχθηκε η δήλωση. Δεν αναφέρθηκε ε, λέξη για τις ε, αποτρόπες δηλώσεις του πρόεδρου Μπασίρ που απείλησε να κόψει τις ε, γλώσσες και τα δάχτυλα των διεθνών παρατηρητών. Η ΣΥΠΗ είναι σημαντική και σίγουρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε παρουσία ώστε να μην ε, γίνει και το Νότιο Σουδάν ε, ένα κράτος σαθρό που θα διοικείται από ένα δικτάτορα. Θέλουμε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις ε, και μετάβαση στη δημοκρατία ε, και του Βόρειου Σουδάν και πραγματικά έμεινα εμβρόντιτη με την δήλωση αυτή που δείχνει ότι δεν έχουμε αυτόνομη στρατηγική για το Σουδάν, απλώς είμαστε ουραγοί των Αμερικανών. Και για την Γουινέα Μπισάο, μετά από αυτά που είπατε και αυτά που ακούσαμε χθε από την ε, Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας, αν θέλουμε ε, να κάνουμε τη διαφορά στη Γουινέα Μπισάου, εμείς θα πρέπει να παραμείνουμε εκεί και όχι να αφήσουμε τους Αμερικανούς που θέλουν να μεταβούν και να φροντίσουν να αναλάβουν την κατάσταση στα χέρια τους. Ε, Λίζεκ. Ο κύριος Λίζεκ, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα ήθελα να αναφέρω, αναφερθώ σε ένα θέμα που είναι σημαντικό ε, και γιατί φορά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Πρόκειται για την Γεωργία και τα γενικά συμπεράσματα από τη του Λουξεμβούργου είναι γενικώ δίκαια και κανένας δεν έχει αντιρρήσεις με τα συμπεράσματα αυτά. Άλλωστε νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε η ανάγκη διατήρησης της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακαιρεότητας καθώς και της κυριαρχίας της γεωργίας. Και αυτή η ανεξαρτησία και η κυριαρχία ευτυχώς υπάρχουν. Δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα με την εδαφική ακαιρεότητα της γεωργίας. Ερωτώ λοιπόν κύριε Διευθυντά, θα μπορούσατε να μας δώσετε λίγες πληροφορίες για τη συζήτηση ε, περί της γεωργίας το Συμβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποιες σκέψεις για το πώς θα συνεχίσει τις δράσεις της ώστε να εξασφαλίσει την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας. Γιατί καλώς συνεχίζονται οι συνομιλίες της Γενέβης, αλλά η μόνη τους προστιθέμενη αξία είναι ότι ακριβώς συνεχίζονται, ότι δεν έχουν σταματήσει. Μήπως όμως θα μπορούσαμε να αναλάβουμε επιπλέον δράσεις, ίσως διμερείς συνομιλίες με τη Ρωσία για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Και η τελευταία παρέμβαση της, ε, του κυρίου Μπουτικόφερ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εχθές η Herald Tribune έγραφε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέρχεται στη διάσκεψη για τη μη διάδοση των πυρηνικών, ενώ ήδη έχει αποτύχει να κλείσει το θέμα αυτό στο εσωτερικό της και επικαλείται ως πηγή ανώνυμα κάποιο διπλωμάτη ε, που κατηγορεί ορισμένα κράτη για τις ε, φιλοδοξίες τους ή για έλλειψη μάλλον φιλοδοξιών ως προς το πυρηνικό αφοπλισμό. Εσείς, κύριε Κούπερ, συμφωνείτε με αυτά τα σχόλια. Και δεύτερη ερώτηση στα γερμανικά που αφορά την απόφαση τη σχετική με την Ουκρανία η οποία ε, αντιφάσκει με την ε, συμφωνία για τον στόλο στη Μαύρη Θάλασσα, στον Εύξηνο εμένουμε σε αυτήν την απόφαση. Θεωρούμε ότι είναι καλή, την υποστηρίζουμε ή εκφράζουμε τη λύπη μας γιατί ε, εντείνει τις διαφορές και αυξάνει τις αποστάσεις μεταξύ ημών και Ρώσων και Ουκρανίας. Ή αδιαφορούμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούπερ έχει πέντε λεπτά για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για τις ερωτήσεις κυρίας Γκόμες. Θα ήθελα να απαντήσω ότι το Συμβούλιο τις συζητήσεις του τις έκανε με προοπτική τη CPS στο συνέδριο και όχι αναφερόμενο στο παρελθόν. Εξού και όντως εκφράστηκε με κάπως διπλωματική γλώσσα και όχι με πιο περίφραστους όρους όπως αυτούς που χρησιμοποίησε η κυρία Γκόμες. Παρά τη διαφορά όμως του λόγου, νομίζω ότι δεν διαφωνούμε ως προς την ουσία. Μόνο ο τύπος της εκφράσεως διαφέρει. Επίσης δεν βλέπω μεγάλη διαφορά μεταξύ ημών και ημών ως προς τους στόχους που επιδιώκουμε. Μας ενδιαφέρει το τι θα γίνει στο Νότο μας ενδιαφέρει ο κίνδυνος της εξασίας της βίας και οι διάφορες μορφές που προσλαμβάνει η βία. Και επίσης, ε, για να χρησιμοποιήσω και πάλι διπλωματική ορολογία, ήταν ε, νοθευμένες οι εκλογές στο Σουδάν, ναι. Ωστόσο ήταν θετικό το ότι έγιναν, γιατί δεν είναι καθημερινό φαινόμενο όπως φαντάζεστε και όλες οι αποστολές παρατηρητών έτυχαν πολύ θετική υποδοχής ακόμη και από εκείνα τα κόμματα τα οποία απέσχουν των εκλογών. Άρα το Σουδάν έχει τη βούληση να γυρίσει μια πολιτική αντιπαράθεση, μια πολιτική, ε, ένα πολιτικό διάλογο και όχι Και αυτό είναι σαφές από τις παρατηρήσεις μας εκεί. Επίσης για η Γουινέα Μπισάο επαναθεωρούμε τις ε, θέσεις μας βεβαίως, αλλά δεν μπορώ να πω ότι θα εγκαταλείψουμε τη Γουινέα Μπισάου. Μάλλον θα πρέπει να δούμε τους όρους υπό τους οποίους θα συνεχίσουμε να έχουμε παρουσία εκεί. Για τον κύριο Λίσεκ και τη Γεωργία. Ναι, καταγράφεται στα συμπεράσματα, αν και δεν συζητήθηκε σε επίπεδο συμβουλίου, Βεβαίως και υποστηρίζουμε την εδαφική ακαιρότητα της γεωργίας, στασόμεθα ως βασική αρχή υπέρ της εδαφικής ακαιρότητας της γεωργίας. Δεν είναι ένα ζήτημα στο οποίο μπορεί να αναπτύσσεται κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις στην ε, Γενέβη σας στόχο έχουν μάλλον να βελτιώσουν τη σταθερότητα στην περιοχή και χάρη σε αυτές τις ε, συνομιλίες εξασφαλίσαμε από τις άλλες πλευρές και κυρίως τους Ρώσους να χειρίζονται κατά διαφορετικό τρόπο τα ε, διάφορα μικροεπισόδια. Στόχος δηλαδή είναι η σταθερότητα, η ασφάλεια των ε, τοπιών πληθυσμών, η, ένα, η επικράτηση ήρεμου κλίματος και στη συνέχεια όταν εξασφαλίσουμε αυτά μπορούμε να συζητήσουμε τα πολιτικά ζητήματα που ενδεχομένως να θέσουν και ζήτημα εδαφικής ακαιρεότητας. Ε, μέχρι τότε όμως έχουμε πολλή δουλειά. Και φυσικά στις συνομιλίες της Γενέβης πρέπει να πω συμμετέχουν και οι Ρώσοι. Ναι και όντω είναι ένα ζήτημα η γεωργία το οποίο θίξαμε, έφυξε η κυρία Άστον ε, όταν επισκεφθεί τη Ρώσα πρόσφατα. Το θίγουμε δηλαδή σε κάθε περίπτωση σε συνομιλίε με του Ρώσου για τον κύριο για την συνθήκη περιμή διάδοσης των πυρηνικών. Το Συμβούλιο το ίδιο δεν ασχολείται με ζητήματα αριθμού πυρηνικών κεφαλών που διαθέτει κάθε χώρα. αλλά νομίζω ότι με μια γενική εικόνα που έχουμε από τα ευρωπαϊκά κράτη, ο αριθμός των πυρηνικών κεφαλών που κατέχουν, που διατηρούν, είναι ελάχιστος. Είναι τόσο χαμηλός που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναφέρεται στο ελάχιστο επίπεδο αποτροπής. Και το Συμβούλιο επεξεργάζεται στη συζήτηση του όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, συνθήκη περί διάδοση, δηλαδή και την διάδοση και, την, ε, και τον πυρηνικό αφοπλισμό και την ασφάλεια. Για δε την Ουκρανία, είναι ένα θέμα ύψης της προτεραιότητας, θα μας απασχολήσει και στο μέλλον ασφαλώς. Βέβαια είναι κυρίαρχο κράτος η Ουκρανία και θα πρέπει μόνη της να αποφασίσει το πώς θα χειρίζεται τη σχέση της με τη Ρωσία. Εμείς δεν θεωρήσαμε ποτέ όταν δική μας δουλειά να αποκολλήσουμε την Ουκρανία από τη Ρωσία. Είναι χώρα όμορη με την Ρωσία και είναι αυτονόητο και αναπόφευκτο να έχει στενές σχέσεις με αυτήν. Δεν έχουμε δηλαδή ανταγωνιστική σχέση με τη Ρωσία εμείς. Και όπως είπα, η Ουκρανική κυβέρνηση είναι εκείνη η οποία θα αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσει τους, τις σχέσεις με τη Ρωσία. Αλλά και πάλι είναι ένα θέμα το οποίο δεν συζητήθηκε στο Συμβούλιο, μάλλον θα τους απασχολήσει το προσεχές στο εγγύς Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε δόκτωρα Κούπερ για τη συνεργασία σας και για την συνεισφορά σας στον εμπαθημένο διάλογο σας. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην εργασία σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Περνάμε στο επόμενο θέμα της μερίσιας διάταξης, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα έφτασε σε πολιτική συμφωνία ως προς το κείμενο ε, στο οποίο αποφάσισε, ε, το οποίο αποφασίστηκε υπό την ε, ύπατη εκπρόσωπο. Και ανοίγει ο δρόμος για τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σύσταση αυτής της υπηρεσίας. Θα ήταν λοιπόν ε, σκόπιμο ο κύριος Μπρόκ και σύμφωνα με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων υπό τον κύριο Βερχόφστατ να προβάλλουμε συγκεκριμένες τροπολογίες σε σχέση με τις γενικές αρχές που διέπουν αυτό το non-paper. Σήμερα περνάμε σε μία νέα φάση διαβουλεύσεων για αυτό το σημαντικό θέμα. Δίνω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Μπροκ, για να, μας, ε, να αποτιμήσει την κατάσταση ως προς τη βασική συμφωνία, καθώς και τα βασικά σημεία του εγγράφου εργασίας που έχετε όλοι. Κύριε Μπρόκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το έγγραφο που έχετε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι όμως έγγραφο εργασίας που μπορεί να πάσα στιγμή να τροποποιηθεί και εξ αρχής σας καλώ να μας δώσετε προτάσεις σε όποιο σημείο βλέπετε ότι έχετε κάτι να προσθέσετε, να τις επεξεργαστούμε εγκαίρως, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταθέσουμε στη συνέχεια την έκθεση, το έγγραφο αυτό εργασίας ως έκθεση. Θα σας εξηγήσω το έγγραφο λοιπόν αυτό πιο συγκεκριμένα, γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για το, να έχουμε τον κανονισμό για το προσωπικό ως σύνολο. Είναι με ένα σύνολο, αλλά πρόκειται ουσιαστικά για 4 ή 5 διαφορετικά έγγραφα και θα πρέπει να δούμε, να ξεχωρίσουμε σε ποιο έγγραφο θα γράψουμε, θα περιλάβουμε τι. Και γι' αυτό, ανεξαρτήτως των όσων περιλαμβάνονται στο έγγραφο για τις αποφάσεις του Συμβουλίου, την κοινή θέση του Συμβουλίου για την ε, διαπραγμάτευση, γιατί πέραν αυτού δεν υπάρχει τίποτε άλλο, δεν είναι δηλαδή μια επίσημη απόφαση του Συμβούλιο. Θα πρέπει εμείς να δούμε τι θέλουμε να αλλάξουμε από το κείμενο αυτό για τα πέραν του Συμβουλίου και τι άλλο θέλουμε να προσθέσουμε. Και να σας πω γιατί. Έχουμε λοιπόν μια διαδικασία διαβουλεύσεως. Και το Συμβούλιο μπορεί βεβαίως να την τροποποιήσει. Όταν έχουμε λοιπόν διαδικασία συναπόφασης για τον κανονισμό το σχετικό με το προσωπικό και διαπιστώνουμε ότι ουσιώδη ζητήματα καθοριστικής σημασίας για τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου και τον προπολογισμό και την απαλλαγή πρέπει να ε, προσδοριστούν έτσι ώστε να έχουμε και στο μέλλον τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τα, τις εξουσίες για τη συναπόφαση. Για να μην ε, διαπιστώσουμε όταν έρθει η ώρα για την αναθεώρηση το 2013 ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει εις βάρος μας και ότι έχουμε χάσει εξουσίες μας. Και γι' αυτό λοιπόν στο άρθρο 6 της, του εγγράφου όπου γίνονται οι προτάσεις για τις τροποποίησεις στη, στα σπέσματα του Συμβουλίου έχουμε και σε συνεννόηση με τον ε, συνάδελφο Ράπκαη πει ότι αυτό θα πρέπει να περιληφθεί στον κανονισμό για το προσωπικό και όχι στις, ε, στα του Συμβουλίου. Σε αυτό, στα, στον κανονισμό θα πρέπει να υπαχθεί. Απόφαση του Συμβουλίου. η συμφωνία σε επίπεδο συμβουλίου δεν αποτελεί για μα, πιστεύω, βάση διαπραγμάτευση, έστω και αν μπορεί να μα καθοδηγήσει, να μα δώσει σωστέ κατευθύνσει, αλλά δεν ε, λύνει κάθε πρόβλημα. Στην πρόταση που σα έχουμε υποβάλει, την προσωρινή αυτή πρόταση, έχει ε, συμπεριληφθεί, έχει ληφθεί υπόψη ε, η τοποθέτηση του Συμβουλίου. Δηλαδή, ό,τι θεωρήσαμε καλό από αυτήν, το έχουμε συμπεριλάβει. και έχουμε επισήμως αναφερθεί και στην τροποποίηση του εγγράφου Άστον και στα όσα έχουν συζητηθεί σε επίπεδο Συμβουλίου. Και επίσης έχουμε, όπως και στο παρελθόν, μια καθοριστική διαφορά, η οποία είναι πως θα πρέπει να είναι προσκολλημένη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο σε δημοσιονομικό και οργανωτικό η υπηρεσία αυτή της εξωτερικών σχέσεων, εξωτερικής δράσης και επίσης λέμε ότι ο διοικητικός του προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι τμήμα του τμήματος 3 και όχι ένα νέο 6. Ταυτόχρονα λέμε και πολύ ξεκάθαρα ότι δια, διαφαίνεται ο generis χαρακτήρας αυτής της υπηρεσίας, ο οποίος συνεπάγεται ότι τόσο για το προσωπικό όσο και για τον προϋπολογισμό ότι θα πρέπει να ε, έχουμε λύσεις κατάλληλες ε, που να εξυπηρετούν ε, το ρόλο αυτών και οι οποίες θα πρέπει να ενσωματώνουν και τις ε, ανάγκες, να ενσωματώνουν τις πτυχές που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες του Συμβουλίου περισσότερο και των δράσεων του Συμβουλίου, όχι μόνο της Επιτροπής. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν είμαστε διατεθειμένοι να επιμένουμε έτσι ώστε τα ζητήματα και τα δημοσιονομικά της ε, αρμοδιότητας του, των αρμοδιότητων του Κοινοβουλίου να διαφυλαχθούν και να επιληθούν κατά τρόπον ουσιαστικό και αποτελεσματικό. Με βεβαίως την υπαγωγή στον έλεγχο από την Όλαφ, αλλά ταυτόχρονα και με διαφύλαξη των ε, προνομιών του Κοινοβουλίου. Επομένως, χρειαζόμαστε επαρκής εγγύηση από πλευρά του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Μέχρι τώρα δεν τις έχουμε δει. Σε αυτό θα κρυθούν πολλά άλλα πράγματα. και για τον, δημοσιονομικό, για τον κανονισμό του σχετικό με το, με το προσωπικό καθιστούμε σαφές ότι πρέπει να υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις πίστεως για το προσωπικό, αφοσίωσης δηλαδή, αυτό το οποίο αναφέρουμε στο άρθρο 9 ως ε, δραστηριοποίηση του προσωπικού της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, εάν στην πλειονότητά του. Το προσωπικό της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης είναι διπλωμάτες της Καρκέρας οι οποίοι έρχονται για μερικά χρόνια σε αυτήν για να γυρίσουν μετά στις έδρες τους, δηλαδή στις εθνικές τους υπηρεσίες, μάλλον δεν θα έχουν ως κύριο γνώμονα το συμφερόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα θα πρέπει να υπάρξει κάποιο άλλο μέτρο η δυνατότητα για αυτούς τους ανθρώπους να επιλέξουν να παραμείνουν στην υπηρεσία, φυσικά χωρίς να απολένουν και το δικαίωμα επανόδου στην εθνική υπηρεσία. Αυτά είναι ζητήματα αρχής. Διότι το λέω, διότι έχω μερικές φορές την εντύπωση σε συνομιλίες με εθνικούς ε, διπλωμάτες, μερικές φορές για προσωπικό, ότι, για, με υπουργούς, ότι δηλαδή σε θέματα προσωπικού ε, θεωρούν τους, το προσωπικό που αποστέλουν ως ιδιοκτησία του τα κράτη-μέλη. Και ότι ως εκ τούτου αυτό το προσωπικό πρέπει να αποτελεί και τον φορέα της εθνικής πολιτικής στη θέση που θα αναλάβει σε μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία. Ε, αυτό πρέπει να καταστεί σαφέ λοιπόν, ότι αυτό το προσωπικό, έστω και αν αυτή η υπηρεσία είναι προσαρτημένη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό το προσωπικό έχει καθήκον να επιτελεί ε, το έργο που τον αναθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό είπα ότι εκπρόσωπο έχει διπλό καθήκον και καθοδηγεί την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και αναπτύσσει μια ε, τον συντονισμό μιας ε, μιας ε, ενωμένης κατά κάποιο τρόπο εξωτερικής πολιτικής σε πλευρά των κρατών μελών. Αυτή είναι η διάκριση στην οποία προβαίνει η ίδια η συνθήκη και άρα είναι σαφές ότι αυτή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης δεν ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα και την εξουσία των κρατών μελών και των Υπουργείων Εξωτερικών τους. Αυτό πρέπει να το καταστήσουμε εμείς σαφές με το κείμενό μας. Επίσης πολύ σημαντική είναι η πολιτική εκπροσώπηση. Στη θέση του Συμβουλίου διαπιστώνω ότι ο ρόλος του Γενικού Γραμματέως δεν προβλέπεται πλέον κατά τρόπο τόσο πολιτικό όσο αρχικά είχε προβλεφθεί. Αλλά μάλλον ε, διοικητικά καθήκοντα θα αναλάβει αυτός. Και αν κατάλαβα καλά τα λόγια του κυρίου Κριστόφερσον από κάποια άλλη συζήτηση, είχε πει ο κύριος Κριστόφερσον ότι σε περίπτωση απουσίας ή του είπα του εκπροσώπου μπορεί να υπάρξει αντικατάσταση από επιτρόπους για εκπροσώπηση κοινοβούλια και άλλους τόπους. Αυτό βγαίνει ως συμπέρασμα και από το έγγραφο Φερχόφστοτ. Βλέπουμε από την άλλη ότι από το Συμβούλιο ακούγονται διάφορε συζητήσει για το τι θα γίνει σε περίπτωση καθαρός, ζητημάτων καθαρό εξωτερική πολιτική, όπου δεν μπορεί κανεί να αντικαταστήσει τον είπα το εκπρόσωπο και τι θα γίνει εάν πρέπει κάποιο ε, ε, επίτροπο να αναλάβει τέτοιου είδου καθήκοντα ω αντικαταστάτη κτλ. Και είπε και ο ε, ο μου εδώ δίπλα ότι από τα όσα είπε ο κύριος Κούπερ που μόλις ακούσαμε, από ρέι το συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε πολιτική εκπροσώπηση πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Πιτικόφερ θα θεωρούσε σκόπιμη την ανάθεση τέτοιου είδους εξουσιών και καθηκόντων ή αν θα τις θεωρούσε και επαρκής ίσως, αλλά πάντως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε και πάντως αυτό εννοούμε όταν λέμε πρέπει να προχωρήσουμε, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτήν την υπόθεση συνεργασία σε πολιτικό επίπεδο και συνεργασία της κυρίας Άστον ε, σε ρόλο συντονισμού, πολιτικού συντονισμού. Ώστε να μιλάμε με την ίδια φωνή, να ακολουθούμε τους ίδιους, τις ίδιες επιλογές λίγο πολύ στα ίδια θέματα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως βεβαίως και η εφαρμογή και η εκτέλεση επίπεδο επιτροπής αλλά πάνω απ' όλα συνεργασία υπό την καθοδήγηση με κοινέ προτάσεις από τον Επίτροπο, από την Υπατή Εκπρόσωπο. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται και στον τομέα της πολιτικής ετονία, αλλά και στους άλλους τομείς εξωτερικής πολιτικής. Θέλουμε νέο προπολογισμό επίση. Το σε θέση. και γι' αυτό θα ήθελα και να ακούσω προτάσεις τι εννοούμε ως νέο προπολογισμό. Στο Συμβούλιο λένε ότι θα πρέπει να είναι ουδέτερος ω προ τον προπολογισμό, ο προπολογισμό ο σχετικός, ουδέτερη ε, με, ως τον προπολογισμό η επάνδρωση τη υπηρεσία. Ναι, αλλά πώ θα γίνει όταν... Ε, προέρχεται το προσωπικό σε τόσο μεγάλο βαθμό από τα κράτη-μέλη. Και από την άλλη θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι όλο το προσωπικό αμείβεται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και όχι από τους εθνικούς. Αυτό πρέπει να είναι απόλυτα σαφές, ανεκτώτως από πού προέρχεται το προσωπικό της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. δεν θα έχουμε σε τέτοια έκταση το φαινόμενο των αποσπασθέντων που είχαμε στο παρελθόν. Ε, γιατί θα έχουμε το 1 τρίτο του διπλωματικού προσωπικού που θα πρόκειται από τα κράτη-μέλη, το 1 τρίτο που θα είναι στρατιωτικό και μετά κάποιοι άλλοι που θα είναι υψηλού επίπεδου από τα εθνικά Υπουργεία των Εξωτερικών που δεν θα αμείβονται ενδεχομένω, εν πάση περιπτώσει όμω θα έχουν παρουσία κτλ. Ε, ας μην είναι τελείως έξω από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας μην, είναι τελείως, ας μην έχει τελείως εγκαταλείψει τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η υπηρεσία με τέτοιο προσωπικό. Θέλουμε δηλαδή αυτοί που θα δουλεύουν εκεί, ναι, να προέρχονται από τα κράτη-μέλη, αλλά να υπηρετούν. Με βάση βέβαια και την ε, κατανομή τη γεωγραφική και την κατανομή σε φύλλα, τις αρχές και τις ανάγκες, τις προτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να έχουμε μια πολιτική συντονισμένη, μια συνεπή πολιτική και ένα μέσον υποστήριξη και τη ανάπτυξη. Αυτό το έχουμε συζητήσει σε συνεργασία με του συναδέλφου από την Επιτροπή Ανάπτυξη. Έτσι ώστε όπου χρειάζεται να κατατεθούν σχετικές τροπολογίες. Σημαντικό επίσης είναι τα μέσα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 8 να μένουν σε αρμοδιότητες των εθνικών πολιτικών ως προς την ε, λήψη των σχετικών αποφάσεων. Αυτά τα μέσα τα οποία λίγο πολύ καλύπτει και η πρόταση Άστον πέραν του λεγόμενου ε, μέσου σταθερότητας. αν και θα πρέπει να συζητήσουμε στην περίπτωση της διαχείρισης στρατιωτικού και μη στρατιωτικού ε, προσωπικού και ανάληψης δράσης τι είδου συντονιστικό ρόλο θα διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει νομίζω να προσέχουμε τα ιδιαίτερα μελήματα των κρατών μελών σε θέματα στρατιωτικά να γίνονται σεβαστά. Να μην ξεπερνάμε δηλαδή κάποια όρια. και να διατηρούμε μεν την ευελιξία μας ταυτόχρονα γνωρίζοντας ότι μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα πως δεν θα πατήσει κανείς στα, χωράφια, στα στρατιωτικά χωράφια κάποιου άλλου σε επίπεδο συμβουλίου στις τελικές αποφάσεις. Πολλές φορές όταν έχουμε διαχείριση κρίσεων διαπιστώνουμε σε τελική φάση ότι δεν είναι τόσο στρατιωτική η αναστρατιωτική και οι ανάγκες, δηλαδή αποστολής προσωπικού και υλικού, αλλά μάλλον ε, επιμελητιακού χαρακτήρα, όπως είδαμε με την ε, περίπτωση της Ταϊτής. Εκεί ίσως τα πράγματα αλλάζουν και έχουν διαφορετική εκτίμηση τα ζητήματα της, ε, του συντονισμού μεταξύ στρατιωτικής και μη δράσης. Σημαντικό σημείο και τελευταίο από αυτά που θέλω να αναφέρω είναι το 4 ή 5, ο πολιτικός έλεγχος. Οι βασικές αρχές που προβλέπονται στη συνθήκη ουσιαστικά έχουν και εδώ θέση. Αλλά ο πολλαπλασιασμός των ε, ε, συνθήκων ή διατάξεων πολιτικού ελέγχου. Ποιος, πότε, πού είναι υπόλεγος, ποιος ελέγχει, ποιος λαμβάνει αποφάσεις, ε, τι γίνεται με τα απόρριτα έγγραφα, το διπλωματικό προσωπικό, το συμβούλιο, τι τους αποφάσεις παίρνει. Όλα αυτά τα ζητήματα νομίζω μπορούμε να τα υπαγάγουμε και στην ε, θελοντική, στην συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. με την δέσμευση την προφορική που είχαμε ότι θα συζητούνται όποτε χρειάζεται αυτά τα ζητήματα και βεβαίω θα πρέπει να έχουμε και εμεί μια βεβαίωση για το πότε θα ζητηθεί η γνώμη μα σε περίπτωση αποστολών ε, προσωπικού ή υλικού όπου χρειάζεται δηλαδή να δοθεί ειδική εντολή. Νομίζω ότι μπορούμε να στηριχθούμε σε ένα memorandum of understanding ε, για συνεργασία με την, με την υπηρεσία της κυρίας Άστον. Και βέβαια η δυσμενής θέση στην οποία βρισκόμαστε είναι ότι εμείς ως όργανο στο οποίο επικρατεί απόλυτη διαφάνεια πάντοτε έχουμε συνεδριάσει ανοιχτέ τις οποίες μπορεί να συμμετέχει, να συμμετέχει μάλλον τις οποίες μπορεί να παρακολουθεί το Συμβούλιο αλλά δεν μπορούμε ποτέ να συμμετέχουμε εμείς ή να παρακολουθούμε τις συνομιλίες επί του Συμβουλίου. Εκεί πέρα έχουμε μειονέκτημα. Ω εκ τούτου λοιπόν αυτό θα έπρεπε να το επανεξετάσουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσεως για να μπορούμε να παρακολουθούμε τα πράγματα και για να μπορούμε να δώσουμε την έγκρισή μας σε σε κανονισμού του Συμβουλίου. Γιατί αν υπάρξει κανονισμό του Συμβουλίου στον οποίο εμείς δεν με τον οποίο εμεί δεν είμαστε σύμφωνοι ή αν δεν θέλουμε να δώσουμε την ε, έγκρισή μα εκ των υστέρων σε περίπτωση συναπόφαση, έχετε σαφή εικόνα μια σειρά εξαρτήσεων υπαγωγών και όρων, εφόσον συμβεί αυτό δεν θα συμβεί εκείνο και ούτε καθεξής, που πιστεύω χάρη στη νέα συνθήκη θα πείσουν το Συμβουλίο να, κοιτάξουν, να κοιτάξει λίγο διαφορετικά τη συμπεριφορά του στην υπόθεση αυτή και να σταματήσει να θέτει προσκόμματα στην ενημέρωση τη δική μας στα θέματα της εξωτερικής δράσης. Ευχαριστώ πολύ. Grazie, collega ε, Ως προς τη σειρά των παρεμβάσεων, καταρχήν με τον κύριο Φερχόφστατ, που είναι εισηγητής από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, μετά η Σκιώδης, και όλοι όσοι ζητήσουν το λόγο στη συνέχεια. Ε, δίνω το λόγο στον κύριο Βερχόφστατ και σας υπενθυμίζω ότι επειδή πολλοί ζήτησαν το λόγο, θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί προς το χρόνο. Δεν μπορούν παρεμβάσεις να υπερβούν τα δύο λεπτά. Δεν θέλω να χτυπάω το σφυράκι, είναι άκρος αντιπαθητικό. Μην με αναγκάστε να το κάνω. Καταρχήν, θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτά που προείπε ο κύριος Μπροκ. Ξέρετε ότι είναι οι ίδιες τροπολογίες οι οποίες υποβλήθηκαν εδώ, υποβάλλονται εδώ που υποβλήθηκαν και στη δική μας Επιτροπή, την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Αυτό έγινε σήμερα το πρωί και μπορώ να σας πω ότι η αντίδραση ήταν γενικά θετική ως προς τις τροπολογίες του κυρίου Μπρόκ και τις δικές μου στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Επίσης, κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία, στις τροπολογίες αυτές θα υπογραμμίσω την συνοχή της εξωτερικής πολιτικής που εγγυούμαστε με αυτές τροπολογίες. Ως προς την Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας, εμείς μεταβήκαμε στην Επιτροπή, είπαμε θα πρέπει να υπάρχει μια συνεκτική πολιτική και να μην κάνουμε αυτό που έγινε με την, να μην γίνει αυτό που έγινε με την πρόταση του Συμβουλίου, δηλαδή τα οριζόντια θέματα αφορούν την Επιτροπή και όταν πρόκειται για γεωγραφικά ζητήματα, έχουμε τις εξωτερικές υποθέσεις, όσον αφορά την ε, εφαρμογή επανερχόμαστε στην Επιτροπή. Όχι, αυτό το αποφεύγουμε με τις τροπολογίες, οδηγούμαστε σε μία απλούστευση. Εξωτερικές υποθέσεις για τον προγραμματισμό, εφαρμογή υπηρεσίες της Επιτροπής, διότι υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος μεταξύ Κομισιών, και ε, υπηρεσίες εξωτερικών υποθέσεων. Αυτή είναι, αυτό είναι το φιλοσοφικό υπόβαθρο που διέπει τις τροπολογίες. Γι' αυτό ακριβώς ε, προτείνουμε και λέμε ότι αποτελεί μέρος του τμήματος 3 του προϋπολογισμού. Δηλαδή, του πιο σημαντικού τμήματος του προϋπολογισμού που σχετίζεται με την ε, Επιτροπή. Και τέλος, ε, κύριε Πρόεδρε, Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε άλλες ε, τροπολογίες που ίσως καταστούν αναγκαίες σε σχέση με αυτές που συντάξαμε μέχρι τώρα, διότι αν το Συμβούλιο δεν κινηθεί προς την κατεύθυνση που επιθυμούμε, εγώ σας λέω ότι είμαι της γνώμης ότι θα χρειαστούμε άλλες ε, τροπολογίες όπου θα επανέλθουν όλες οι κοινοτικέ αρμοδιότητες της Επιτροπής προς την Επιτροπή. Θα έχουμε επαναφορά αρμοδιοτήτων δηλαδή. Εάν λοιπόν χρειαστούν άλλες επιπρόσθετες τροπολογίες. Όλα βεβαίως θα εξαρτηθούν από την αντίδραση του Συμβουλίου προς τις ε, δικές μας τροπολογίες που υποβάλλονται σήμερα. Άρα ίσως θα επανέλθουμε με άλλες ε, τροπολογίες για να επανέλθουν πολλές αρμοδιότητες, συνεργασία, πολιτική γειτονίες, να επανέλθουν στην Επιτροπή. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια υπηρεσία εξωτερικής δράσης και να την ε, χρησιμοποιήσουμε για να αδειάσουμε την ε, κοινοτική μέθοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό αποφεύγουμε με τις τροπολογίες μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη έχει το λόγο. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ε, οι τροπολογίες έχουν, ε, μας δίνουν μια θετική τροπή ως προς το έγγραφο της ΥΠΑ της εκπροσώπου πρόκειται για ένα ε, οργανικό έγγραφο το οποίο προβάλλει τις θέσεις μας των τελευταίων εβδομάδων. Ως εισηγητών η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, είχε μία πραγματιστική προσέγγιση που ξεκινά από αρχές και όχι διατυπώσεις, δηλαδή πλήρη έλεγχο του Κοινοβουλίου, συνοχή, εξωτερική δράση και μία γεφύρωση μεταξύ κοινοτικής πολιτικής και διακυβερνητικής. Εγγυόμενη την κοινοτική πολιτική, ιδιαίτερα όσον αφορά το αναπτυξιακό σκέλος βάζω κατά μέρος το οντολογικό θέμα του ε, οργανογράμματος της υπηρεσίας. Ως προς τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, νομίζω ότι το έγγραφο περιλαμβάνει πολλά βασικά ε, ζητήματα. Μερικά από αυτά ανατέθηκαν στις ε, επιπρόσθετες συμφωνίες θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα των ακροάσεων στο Κοινοβούλιο, να το δούμε με τους επικεφαλείς αντιπροσωπιών και τους αξιωματούχους της υπηρεσίας. Επίσης είναι ύψης της σημασίας η αναθεώρηση της διαθεσμικής ε, συμφωνίας ε, ως προς το ως προς την ΚΕΠΑ, διότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να δούμε τι αρμοδιότητες μπορεί να έχει το Κοινοβούλιο στον τομέα της κοινή εξωτερικής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Ως προς το κοινοτικό σκέλος, το έγγραφο μας δίνει μία επιλογή, μία εναλλακτική σε σχέση με τις υπηρεσίες της ε, αυτές και τις αρμοδιότητες που ενέπιπταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι ε, ο ρόλος που ανατίθεται στην υπηρεσία είναι πολύ ψηλό σε σχέση με τους επιτρόπους ανάπτυξης. Πρόκειται για κάτι το διαφορετικό από αυτό που ζήτησε ο κύριος Φερχόφστατ, δηλαδή μια διαφορετική ε, ρύθμιση μεταξύ Κομισιών και Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Αυτό το θέμα θα πρέπει να το εμβαθύνουμε ήδη από τώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γκραφ Λάμστορφ ε, από τους Φιλελεύθερους. Πρόεδρε, ευχαριστώ με πολύ ενδιαφέρον διάβασα το έγγραφο των δύο συναδέλφων. Είναι πολλά σημαντικά στοιχεία αυτά τα που έχουν περιλάβει στο κείμενο. Είναι σημαντικό ιδιαίτερο στο Κοινοβούλιο να έχει τη θέση του στη λήψη αποφάσεων και να υπενθυμίσει στα άλλα όργανα τη θέση του αυτή. Στον πυρήνα της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης είναι η διαχείριση των κρίσεων, το στρατιωτικό δηλαδή σκέλος και η συμπερίληψη του πολιτικού σκέλους και του σκέλους της ασφάλειας. Είναι σωστή λοιπόν η κατεύθυνση στην οποία ακολουθεί το έγγραφο. Βέβαια κάποιες λεπτομέρειες θα πρέπει να ε, ρυθμιστούν, αλλά πάντως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η, ε, του προσωπικού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη του προσωπικού και δι του στρατιωτικού προσωπικού, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε προβλήματα ε, σχετικά με, τις, ε, με το ρόλο του προσωπικού, στρατιωτικού προσωπικού ή του πολιτικού προσωπικού που διαχειρίζεται κρίση στην υπηρεσία εξωτερική δράση. Και γι' αυτό νομίζω θα πρέπει να γίνει διασύνδεση με τον ε, κανονισμό προσωπικού. Επίσης, η εκπροσώπηση, και συμφωνώ με τον κύριο Μπροκ, από το Κοινοβούλιο έχει κάπως μετακυλήσει τις αρμοδιότητες ε, μεταξύ των δύο αυτών θεσμών, δηλαδή δεν εντοπίζονται όλες οι αρμοδιότητες εκπροσώπησης στον Γενικό Γραμματέα. Ίσως θα πρέπει να δούμε αν ο Γενικός Γραμματέας θα ονομάζεται στο μέλλον Γενικός Διευθυντής ή αν θα βρεθούν κάποιοι άλλοι ρόλοι για τον Γενικό Γραμματέα. Πάντως το σημαντικό είναι να υπάρχει ένας πολιτικός μηχανισμός συντονισμού. Συντονισμού διαφορετικών πολιτικών παραδόσεων, κουλτούρας ή νοοτροπίας διαφορετικής που θα πρέπει να αναλάβει και βέβαια ο υπατός εκπρόσωπος και ο Γενικός Γραμματέας ή όποιος, όπως ονομάζεται αυτός. για τους πρασίνους η συνάδελφος ε, Λούνατσεκ που αντικαθιστά την κυρία Μπραντνερ. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπροκ γιατί κατάφερε να συμπεριλάβει και μερικές δικές μας παρατηρήσεις για την εξωτερική υπηρεσία. Και προτιμώ την τελευταία εκδοχή του εγγράφου του από την αρχική. Τον ευχαριστώ θερμά για τις αλλαγές. Συμφωνώ με τα περισσότερα που είπε ο κύριος Μπροκ. Θα ήθελα να επισέλθω σε ορισμένες λεπτομέρειες που είναι σημαντικές για μας. Το ένα αφορά την πολιτική εκπροσώπηση. Πολύ σωστά, όπως σας είπε ο κύριος Ντονζόν, κύριε Μπροκ, ενημερωθήκατε για τις παρατηρήσεις του κυρίου Κούπερ. Κάτι που αποδεικνύει ότι χρειαζόμαστε πολιτική εκπροσώπηση. Λυπάμαι που το επαναλαμβάνω, αλλά είναι γεγονός πράγματα σημαντικά για μας. Το θέμα του χρηματοπιστωτικού μηχανισμού είναι σημαντική δυνατότητα αυτή και θα πρέπει να παραμείνει σε όλα τα στάδια στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ σημαντικό. Επίσης δεν έχουν δοθεί απαντήσεις για τις ευθύνες. Δεν ξέρω αν θα μπει στο, στον κανονισμό του προσωπικού, αλλά προς το παρόν παραλείπεται το θέμα αυτό. Και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χαιρόμαστε ότι αποσαφηνίστηκε ότι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι κεντρικά σημεία όλων των αντιπροσωπιών. Στο κείμενο του Συμβουλίου όμως δεν αναφέρεται σαφώς αυτό. Θα πρέπει να διευκρινιστεί λοιπόν τι θέματα ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ε, αναφέρονται εδώ. Θα είναι μονάδα, θα είναι ε, γενική διεύθυνση, γιατί αν θέλουμε να δώσουμε κεντρικό χαρακτήρα στα ανθρώπινα δικαιώματα και, τις, ε, και τη δημοκρατία θα πρέπει να έχουμε ειδική διεύθυνση γι' αυτό. Επίσης, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, είπαμε, θα είναι ανοιχτή από εκπροσώπους ε, των ε, Υπουργείων, όχι μόνο όμως από τις διπλωματικές υπηρεσίες, αλλά και από εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξη, για παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σε ό,τι αφορά το φύλλο, την ισορροπία μεταξύ των φύλων, χαίρομαι που αναφέρεται αυτό για το προσωπικό, αλλά γιατί να μην αναφέρεται γενικώ στην, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράσης αυτό το θέμα τη εισεκπροσώπησης των φίλων, Εκ μέρους τη ε, της ΓΚΟΕ, κύριο Σούλτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και στην Επιτροπή συνταγματικών ε, υποθέσεων είχα την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον κύριο Φερχόφσταφ για την πολύ καλή συνεργασία και τώρα να ευχαριστώ και τον κύριο Μπροκ. Έχουμε να κάνουμε εδώ με το interfacing, δηλαδή την συνεργασία στα θέματα που ανήκουν πραγματικά στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και εκείνων των θεμάτων τα οποία δεν ανήκουν αποκλειστικά στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης όπως εξωτερικό εμπόριο κτλ. Και εδώ στην Επιτροπή μας, θα έπρεπε να επισημάνω ακόμη μία πτυχή η οποία δεν είναι τόσο ξεκάθαρα νομίζω καταγεγραμμένη στην έκθεση των ε, δύο συναδέλφων και αναφέρομαι στην πολιτική πρόληψη των συγκρούσεων. Εδώ βλέπω δύο χωριστά. Ε, ε υπήρχαν μάλλον μέχρι τώρα δύο χωριστά κεφάλαια. Ένα για την πολιτική Υποτροπή και ένα για τη στρατιωτική. Ε, τώρα είναι συνδυασμένοι τα δύο σκέλη, όμως δεν βλέπουμε στην πρόληψη των συγκρούσεων ποιο είναι αρμόδιο Αυτό το θυμάμαι μάλιστα από τι συζητήσει που είχαμε κάνει με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή στην κυρία Άστον θα προσφέρουν τι σχετικέ ε, συμβουλέ, ε, οι εκπρόσωποι του στρατιωτικού σκέλου και όχι οι διπλωμάτε, όχι το πολιτικό σκέλο. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα χωριστό τμήμα για την πρόληψη των κρίσεων με την πολιτική διάσταση αφενός και το πολιτικό σκέλο, ε, δηλαδή την ασφάλεια και την άμυνα αφετέρου, το στρατικό σκέλος. η δε αναπτυξιακή πολιτική ίσως θα έπρεπε να αναπτυχθεί περισσότερο. Έχουν γίνει πολλές ανταλλαγές απόψεων, ε, πιστεύω, που ήδη αναφέρθηκαν στη συζήτηση. Αλλά θα ήθελα και να υπογραμμίσω το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να χειριστεί τα θέματα της αναπτυξιακής πολιτικής και να διαφυλάξει τις προνομίες του, γιατί πρόκειται για τομείς τους οποίους δεν μπορούμε να χάσουμε από τις αρμοδιότητες μας. Είναι αισθήματα στην απόφαση και πρέπει να τα διαφυλάξουμε ο κύριος Σαλαφράγκα στη συνέχεια. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους κυρίους Μπροκ και Βερχόφστατ για τα έγγραφά τους. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσουμε ότι η πολιτική απόφαση και η συμφωνία του Συμβουλίου Υπουργών είναι η βάση για τις διαπραγματεύσεις. Και πολύ σωστά ο κύριος Μπροκ είπε ότι θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε για το θέμα αυτό πριν ε, ικανοποιηθούν οι διεκδικήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το σχέδιο απόφαση αναφέρει ότι θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της έγκριση του από το Συμβούλιο. Και μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή του, είπατε εκπρόσωπο θα υποβάλει τι ε, δημοσιονομικέ προτάσει. Νομίζω θα ήταν λάθο να ανοίξουμε όλα μας τα χαρτιά στο μέτρο που έχουμε συναπόφαση για την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού και το, την, το καταστατικό για το προσωπικό, τον εσωτερικό κανονισμό του προσωπικού. Όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Μπρόκ, δεν θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε αν δεν ικανοποιηθούμε πλήρως από το Συμβούλιο ω προς τις διεκδικήσεις μας. Και οι προτάσει των κυρίων Μπρόκ και Φερχόφστατ είναι πολύ συνετέ ό,τι αφορά την πλήρη ε, πολιτική και δημοσιονομική ευθύνη της υπάτης εκπροσώπου θα ήθελα να κάνω μια πρόταση. Ό,τι αφορά το μηχανισμό πολιτικού συντονισμού, στην παράγραφο 2β, ίσως ήταν ενδιαφέρον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εντάξει αυτό το μηχανισμό πολιτικού συντονισμού. Μεταξύ άλλων, γιατί ήδη ίδια είπατε εκπρόσωπο στην πρότασή τη μα λέει ότι θα έχει διαβουλεύσει και θα στήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τι βασικέ πτυχέ και τα θεμελιώδη σημεία τη εξωτερική πολιτική και θα φροντίσει να ληφθούν όντω υπόψη οι θέσει του Κοινοβουλίου από το Συμβούλιο. Από αυτό το πρίσμα, σκόπιμο θα ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμπεριληφθεί και στον μηχανισμό πολιτικού συντονισμού. Είναι συνετές, επαναλαμβάνω, οι προτάσεις ε, και τάσσονται υπέρ της κοινοτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα σας ευχαριστώ γιατί σεβαστήκατε πρώτα απ' όλα το χρόνο σας, ο κύριος Βόμποντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι όντως πολύ καλό το έγγραφο. Σύντομες παρατηρήσεις και λίγες. Καταρχάς, δεν είμαι πεπισμένο ότι η σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου και είπα του εκπροσώπου θα πρέπει να προσδοριστούν μόνο μέσα σε ένα σε μια βάση θεωρητική, νομίζω θα πρέπει, ε, σε μια βάση μόνο πρακτική, θα πρέπει να ορίσουμε και βασικές αρχές μέσα από το έγγραφο και από εκεί και πέρα τις λεπτομέρειες να τις δούμε στην πορεία. Δεύτερον, είμαι σύμφωνος ε, ως προς την ιδέα της διασύνδεσης και της υπαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους επιτρόπους. Θα τα καταφέρουμε, δεν ξέρω, αλλά πάντως θα είναι ε, σκόπιμο να υπάρχει διασύνδεση με τους επιτρόπους που έχουν την αρμοδιότητα στο κάθε τομέα. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι στο 1β έχω κάποιες αντιρρήσεις, διότι οι επίτροποι είναι μέλη της Επιτροπής. Δεν μπορούν να τεθούν στο ίδιο επίπεδο με τους ε, εκπροσώπους της Άστον, τους deputies δηλαδή. Ναι, βεβαίως μπορούν να αντικαταστήσουν οι Επίτροποι την κυρία Άστον, αλλά έχουν άλλο ρόλο. Ο συντονισμός λοιπόν γίνεται πρώτα σε επίπεδο Άστον και Επιτροπής και Επιτρόπων και μετά το δράση αυτού του συντονισμού μπορεί να υπάρξει ένας εκπρόσωπος της Άστον, αλλά δεν μπορώ να βάλω τον αντικαταστάτη της Άστον, τον υπό εκπρόσωπο σε επίπεδο ισότιμο με τον επίτροπο. Αυτό. Λίγες οι παρατήσεις όπως είπα, αλλά γενικά οι κατευθύνσει του εγγράφου και οι προτάσεις του είναι ε, πολύ καλές και τις υποστηρίζουμε. Απλώς παρακαλώ στο 2β, στο 2β να ξανασυλλογιστούμε λίγο αυτό το σημείο. Για δε την ε, συμμετοχή του Κοινοβουλίου ε, δεν πρέπει να την χάσουμε. Εμείς είμαστε η ελεγκτική αρχή θα πρέπει να είμαστε παρόντες και στο συντονισμό και στον έλεγχο ασφαλώς. Κυρία Χάουταλα. Κυρία για τους πράσινους. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λούνατσεκ ήδη σας μίλησε για τη θέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πρόταση αυτή. Θα ήθελα και εγώ να υπερθεματίσω. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι και το Κοινοβούλιο είναι εξίσου ενωμένο με το Συμβούλιο. Και από την άποψη της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα ήθελα να πω ότι η θέση του ειδικού ε, τμήματος που προτείνουμε για το άρθρο 4 για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να έχει υψηλό επίπεδο. Δεν μας αρκεί αυτό το τμήμα να είναι τμήμα δεύτερης κατηγορίας και να μην φτάνει η φωνή του στα υψηλά κλιμάκια της λήψης των αποφάσεων. Γιατί λοιπόν να μην ενισχύσουμε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες αυτού του τμήματος, ό,τι επίπεδο και να έχει, και να το μετατρέψουμε, να γίνεται, σε μια γενική διεύθυνση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να μην είναι ένα απλό τμήμα. Μέχρι στιγμής ε, ο ύπατο εκπρόσωπος, ε, ο κύριος Σολάνα, εκπροσωπώνται για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από έναν ειδικό απεσταλμένο, ειδικό εκπρόσωπο. Δεν θα θέλαμε ε, να υποβαθμιστεί εδώ η φωνή του εκπροσώπου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και το αρμόδιο τμήμα θα πρέπει να έχει σαφείς και εκπεφρασμένες ε, ευθύνες για θέματα ολοκλήρωσης και συμπερίληψης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πολιτική προς όλες τις χώρες. Ακούγοντας τον κύριο Φερχόφστατ, άρχισα, άρχισα να μεζώνουν τα φίδια. Γιατί είπε ότι οι πολιτικές για κάθε χώρα θα, είναι, θα ανήκουν σε κάθε χώρα και τα οριζόντια θέματα θα τα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς θέλουμε μια οριζόντια λήψη υπόψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η κατάρτιση είναι πολύ σημαντική και θέλουμε να υπάρξει επαρκές προσωπικό για να καταρτιστούν σωστά οι αρμόδιοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα στι αντιπροσωπίε. Ο κύριος Σεβερίν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τους δύο εισηγητές μας που μας παρουσίασαν σήμερα κοινέ θέσεις. Το έγγραφο είναι καλό και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε φάση εκλέπτησης ε, της θέσης μας και αποκριστάλλωσης της που θα καταλήξουν στην ενιαία φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέναντι στα άλλα θεσμικά όργανα. Και νομίζω ότι και στη φάση προγραμματισμού και στη φάση εκτέλεσης ε, υπάρχει συνένεση μεταξύ μας. Θέλουμε έναν μηχανισμό πολιτικού συντονισμού που θα εξασφαλίζει μια συνεπή και συνεκτική θέση για το τι επιθυμούμε να κάνουμε και ποιοι είναι οι στόχοι μας και σε ό,τι αφορά τη διαθεσμική συνεργασία, δηλαδή το συντονισμό μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων που θα διαδραματίσουν κοινό ρόλο, αλλά και υπάρχει και ένας διοικητικό συντονισμός που ίσως θα πρέπει να διευκρινιστεί κάπως για το ρόλο του Γενικού Γραμματέα και το επιτελείο του. Και φυσικά η δημοσιονομική διάσταση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από την ίδια συνέπεια γιατί η συνέπεια και η συνεκτικότητα της δημοσιονομικής διαδικασίας θα φανεί και σε προπαρασκευαστική φάση, σε φάση προγραμματισμού, στην φάση της παρουσίασης του προϋπολογισμού, αλλά και στη φάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες του μηχανισμού, πάντως και ο δημοσιονομικός προγραμματισμός, η παρουσίαση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού θα πρέπει να, είναι, να χαρακτηρίζονται από συνέπεια και συνοχή. Και νομίζω ότι η λέξη κλειδιά είναι η διαφάνεια, η υπευθυνότητα, συνοχή, αποτελεσματικότητα και απόδοση ευθυνών φυσικά. Θέλουμε μια τέτοια ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, θα είναι υπόλογη, αποτελεσματικότητα. Και θα ήθελα να προτείνω μια τροπολογία προς τους κυρίους Μπρό και που ελπίζω να βρει σύμφωνο και τον κύριο Σαλαφράγκα και τον κύριο Σβόμποτε και να είναι χρυσή τομή μεταξύ των δύο. Ευχαριστώ κύριο Σάριος Βόλσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εγκομιάσω τους δύο εισηγητέ για την προσέγγιση τους και χαίρομαι που έχουμε κοινή έκθεση και των δύο επιτροπών, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Συνταγματικής Επιτροπής και ευελπιστώ ότι και οι υπόλοιπε επιτροπέ θα ακολουθήσουν την πολιτική φιλοσοφία τη έκθεση αυτή. Νομίζω ότι έγιναν προσπάθειες για μια ευφύ και συνεπή, συνεκτική προσέγγιση σε ό,τι αφορά μια ισχυρή ευρωπαϊκή υπηρεσία που θα χαρακτηρίζεται από την κοινοτική μέθοδο και θα χαρακτηρίζεται επίσης από ομοιομορφία σε αυτή την sui generis δομή της. Αυτή η κοινοτική δομή σημαίνει ανάμειξη όλων των ε, φορέων και συμμετοχή μεταξύ, συμμετοχή τους. Άρθρο 7C ε, και παράγραφος 6 για τη γεωγραφική κατανομή και τα μέτρα που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Μία ισχυρή Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να χαίρει νομιμοποίησης ε, και να, έχει την... και να δίνει σε όλα τα κράτη-μέλη την αίσθηση της ιδιοκτησίας και μάλιστα να έχει όσο πιο ευρεία βάση γίνεται και να σέβεται τις ευαισθησίες και τις ιδιαιτερότητες των χωρών. Και ευελπιστώ ότι οι πρόσωποι μας στις διαπραγματεύσεις θα δείξουν πυγμή και αποφασιστικότητα ώστε να πριτανεύσει η πολύ σωστή δική μας πολιτική φιλοσοφία στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Λέζινγκ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ο Σμίθος αναφέρθηκε και στα αναπτυξιακά μέσα ήδη. Η έννοια των αναπτυξιακών μέσων έχει και στον τομέα των αναπτυξιακών οργανώσεων συζητηθεί και μόνο η... το γραφείο White Case έχει αναλάβει εντολή να συζητήσει την ανάπτυξη των μέσων αυτών υπό το φως της ε, νέα συνθήκη, συνθήκης Λισαβόνας, οποία, το οποίο δε αυτό γραφείο White Case διαπιστώνει ότι υπάρχει διάρρηξη του, της παλαιάς συμφωνίας λόγω της συνθήκης ε, της Λισαβόνας και δεν ήθελα εδώ να παραθέσω τα λόγια τους, λένε λοιπόν ότι περιορίζεται η συμφωνία αυτή στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο στο τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, η αναπτυξιακή βοήθεια κοίται έξω από την ε, σχετική αυτή πολιτική, για την οποία δεν έχει η υπηρεσία αρμοδιότητες. Και γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η απόφαση, αυτή η πραγματογνωμοσύνη καλύτερα πρέπει να μας απασχολήσει. Πρέπει να την εξετάσουμε για να δούμε πώς θα χειριστούμε τα θέματα της αναπτυξιακής βοήθειας. Αυτό δεν το άκουσα, δεν το λέει κανείς μέχρι τώρα. Και ο αρμόδιος για την ανάπτυξη επίτροπος έχει αρμοδιότητες ε, παρακολούθησης και προγραμματισμού, αλλά όχι πολύ συγκεκριμένες. Ε, υποτίθεται ότι συντονίζει το έργο των αναπτυξιακών ε, δραστηριοτήτων, αλλά οι αναπτυξιακές οργανώσεις φοβούνται ότι ο αρμόδιος για την ανάπτυξη επίτροπος ε, και η ύπατη εκπρόσωπος δεν θα έχουν πολύ σαφώς δια, καθορισμένες αρμοδιότητες και σε περίπτωση διαφωνίας, σε σύγκρουση καθηκόντων θα επικρατεί πάντα η δεύτερη. Ευχαριστώ φέρμα. I'm here. Εγώ είμαι συντονιστής τη Επιτροπής ε, προπολογισμών από τους Σοσιαλιστές. Γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω για τον δημοσιονομικό κανονισμό. Νομίζω ότι φτάνουμε σε μια κοινή συνεννόηση επί του θέματος και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής διότι αναφερθήκατε στη Διαθεσμική Συμφωνία για τα δημοσιονομικά γιατί νομίζω ότι θα πρέπει επίση να αλλάξει Έχω ένα ερώτημα προς τον κύριο Μπρόκ, διότι από όσο άκουσα, είπατε για έναν οργανισμό sui generis εντός της Κομισιόν, αλλά αυτό είναι αντιφατικό. Είτε είναι sui generis, είτε εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε θεωρείται υπηρεσία, agency. Άρα δεν πρέπει να αλλάξει ο δημοσιονομικός κανονισμός. Το θέμα sui generis, αν δηλαδή είναι υπηρεσία sui generis, ε, τότε ε, εμπίπτει στο δημοσιονομικό κανονισμό όπως η Επιτροπή Περιφερειών, Ελεγκτικό Συνέδριο, ΔΕΚ και ούτω καθεξής. Άρα θα πρέπει να αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του δημοσιονομικού κανονισμού και να έχει το, την δική της έκθεση απαλλαγής. Διαφορετικά εντάσσεται στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να επέλθει αλλαγή στην πρώτη παράγραφο του Δημοσιονομικού Κανονισμού. Άρα τι εννοείται. Εννοείται η υπηρεσία Sui Generis που θα έχει το δικό της διοικητικό προϋπολογισμό. Όχι στο τμήμα 3 αλλά στα άλλα τμήματα. Βεβαίως ε, τα λειτουργικά έξοδα εντάσσονται στην Κομισιόν αλλά αυτό που είναι βασικό είναι κατά πόσο πρόκειται για υπηρεσία σου generis με δικό της διοικητικό προπολογισμό ή εντάσσεται στην Κομισιόν. Θα ήθελα να μου το διευκρινίσετε αυτό. Κέλλαν από το ΕΛΚ. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου ως προς τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας Νομίζω ότι οι συνάδελφοι ε, Μπροκ και Φερχόφστατ ε, θεωρούνται, θα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ήταν οι αρχιτέκτονες αυτού του μεγάλου οικοδομήματος της υπηρεσίας, ε, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Και νομίζω ότι πρόκειται για μια σωστή εξυψορόπηση του ρόλου δηλαδή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας σε σχέση με την Κομισιόν και το Συμβούλιο δηλαδή που εντάσσεται από ε, πολιτική και δημοσιονομική πλευρά. Επίσης, θα πρέπει να επέλθει μία γεωγραφική εξισορρόπηση ως προς την υπηρεσία αυτή ε, εξωτερικής δράσης. Και αυτή η διπλωματική γεωγραφική εξισορρόπηση θα πρέπει να οδηγήσει και σε μια επέκταση της υπηρεσία για συμμετοχή ε, εθνικών διπλωματών έτσι ώστε να μπορέσουν να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Αυτό αφορά και τον προπολογισμό. Θα πρέπει να προσδώσουμε τα κατάλληλα μέσα σε αυτή τη διπλωματική υπηρεσία εξωτερικής δράσης και το άλλο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω, το τέταρτο, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, μηχανισμός συντονισμού πολιτικών μέσα στην υπηρεσία αυτή. και να υπάρχει ένα τμήμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και για αντιμετώπιση κέριων σημείων ως προς την εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, συμφωνώ με τη συνάδελφο Χαουτάλα. ότι δηλαδή οι αρχές αυτής της εκπροσώπησης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να έχουν μια πιο συγκεκριμένη μορφή. Αλλά μέχρι τώρα το ε, αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα θετικό και με εξέπληξε Κριστόφερσεν που εκπροσωπεί την ε, ύπατη εκπρόσωπο και μετά θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο Μπροκ. Thank Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και που μου επιτρέπετε να σχολιάσω ορισμένες από τις ε, παρεμβάσεις που ακούσαμε σήμερα το πρωί. Καταρχήν, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ κέριο σημείο της διαδικασίας. Έχουμε μία κοινή θέση του Συμβουλίου και έχουμε επιτρέψει επιτάπητος μία ενοποιημένη έκδοση της θέσης του Κοινοβουλίου για, ως προς ανάγκες υποβολής τροπολογιών. Άρα είμαστε σε ένα στάδιο όπου οι πολιτικές διαπραγματεύσεις μπορούν να αρχίσουν. Και είμαι αρκετά αισιόδοξο ως προς την πολιτική αυτή διαπραγμάτευση. Γνωρίζω και ο κύριος Μπροκ αναφέρθηκε σε αυτό ότι σε ορισμένα σημεία ε, εσείς προβάλλετε αλλαγές που αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές του Συμβουλίου και που δέχεται η υπατή εκπρόσωπος. Και βεβαίως αυτές τις είδαμε και στις άτυπες επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα προχωράμε θετικά. Δεν είμαι απεσιόδοξος λοιπόν ότι εν ευθέτω χρόνο δεν μπορεί να επέλθει μια συμφωνία. Και μιλώ για συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς το περιεχόμενο της βασικής απόφασης. Διότι αν επέλθει συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως προς το βασικό σκέλος της συμφωνίας, δεν κατανοώ γιατί θα πρέπει να κρατήσουμε στάση αναμονής για να τεθεί σε εφαρμογή αυτή η συμφωνία, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή πριν επέλθουν τα άλλα στοιχεία, ιδιαίτερα ως προς τον κανονισμό του προσωπικού. Γιατί ίσως ε, να πρόκειται για μια χρονοπόρα διαδικασία η επάνδρωση του προσωπικού και ο χρόνος είναι ένα βασικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας. Βεβαίως υπάρχουν και διαφορές αλλά για να τις ξεπεράσουμε θα πρέπει να υπάρξει αμοιβαία κατανόηση και να ξέρουμε τι πραγματικά αποζητούμε ως προς την ουσία, πέρα από το θεωρητικό σκέλος. Θα ήθελα να πάρω ως παράδειγμα αυτή τη συζήτηση ως προς το κατά πόσο θεσμικά ε, βρίσκεται υπό την αιγίδα της Κομισιόν κατά πόσο πρόκειται για μια ε, αυτούσια υπηρεσία, μια σουγένερης υπηρεσία. Δεν θα ήθελα να υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς ε, το ότι αν μιλάμε για κοινωνικά ζητήματα θα δράσουμε διαφορετικά από το αν πρόκειται για μια γενική διεύθυνση της Κομισιόν. Η ίδια διαδικασία ισχύει για την ε, προετοιμασία των αποφάσεων μέχρι το Διευθυντήριο της Επιτροπής που θα αποφανθεί συλλογικά. Υπό αυτή την έννοια η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα δρά σαν να επρόκειτο για μια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι θα λειτουργήσει. Το γεγονός όμως ότι ζητάμε μία ανεξαρτησία και αυτονομία σε σχέση με τον προϋπολογισμό και το προσωπικό, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή, αυτός ήταν ο όρος που έθεσε το Συμβούλιο για να δεχτεί μια, ευρύτατη, μια υπηρεσία ευρύτατης δράσης, δηλαδή διαχείριση κρίσεων, στρατιωτικές επιχειρήσεις, εξωτερική δράση. Εάν δεν δεχτούμε μια τέτοια ανεξαρτησία, αυτοδυναμία όσον αφορά το δημοσιονομικό σκέλος και το προσωπικό, τότε δεν εμπίπτουμε σε αυτό τον πολιτικό όρο, σε αυτή την πολιτική συνθήκη που έθεσε το Συμβούλιο. Αλλά δεν κατανοώ και το εξής. λέμε ότι εάν ο προϋπολογισμός μας ενταχθεί στο τμήμα 3 του προϋπολογισμού θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια από το αν είναι ένα διαφορετικό ε, τμήμα. Νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια εάν έχουμε τον δικό μας προϋπολογισμό σε ένα διαφορετικό τμήμα. Εδώ μιλώ για τον ε, προϋπολογισμό διοικητικών εξόδων. Εάν έχουμε διαφορετικό τμήμα, υπάρχει πλήρης διαφάνεια ως προς το προσωπικό που εντάσσεται στην υπηρεσία αυτή. Εάν εντάσσεται στον προϋπολογισμό της Κομισιόν, Ε, τότε διαχέεται στο γενικότερο προϋπολογισμό. Άρα δεν μπορείτε να επιδράσετε στον έλεγχο του προϋπολογισμού. Εσείς είσαστε το ένα σκέλος της δημοσιονομικής αρχής, της αρχής επί του προϋπολογισμού και θα έχετε διαφορετική επιρροή αν έχετε να κάνετε με ένα ξεχωριστό προϋπολογισμό παρά αν ενταχθούμε στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή επίσης στο εξής. Είπατε ότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης εντάσσεται στον οργανισμό της Κομισιόν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα έχουμε πολύ ε, προσωπικό, στρατιωτικό προσωπικό, που θα, θα εντάσσονται σε ένα ειδικό καθεστώς. Θα υπάρχουν και εθνικοί διπλωμάτες και ίσως θα ήταν ε, πολύ αρνητικό προηγούμενο εάν θεωρηθεί ε, αυτό το προσωπικό, ένα, ένα κανονικό προσωπικό, το κανονικό προσωπικό που εντάσσεται στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και βεβαίως το προσωπικό, ένα μεγάλο μέρος θα προέλθει από την Κομισιόν ως προς την εκπόνηση των πολιτικών ε, θα προέλθει το προσωπικό από την Κομισιόν περίπου 680 άτομα από τις Βρυξέλλες και από το εξωτερικό 150 από τη γραμματεία του Συμβουλίου από την άλλη πλευρά. Άρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η Κομισιόν δεσπόζει. Ε, υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, αλλά δεν έχω χρόνο να επεκταθώ. Ο κύριος Μπροκ, να, για να σχολιάσει αυτές τις παρατηρήσεις και ό,τι προακούσαμε. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον κύριο Κριστόφερσον που επισήμανε που υπάρχει δυνατότητα για ανοίγματα, για πρόοδο και για επικοδομητική συνεργασία τις επόμενες εβδομάδες. Ας μην υποτιμώ όμως και το Συμβούλιο. Είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε επαρκή σαφήνεια στο τμήμα 3. Δεν χρειαζόμαστε έξωθεν ευλογίες. Και θα τα καταφέρουμε. Εάν πρόκειται να γίνει αυτό αργότερα με τον κανονισμό για το προσωπικό, ίσω χρειάζεται περισσότερη πυθό, προσπάθεια πυθό. αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα καταφέρουμε. Και επιτρέψτε μου να μην ε, απαντήσω διεξοδικά σε όλες τις παρατηρήσεις. Ε, θα αναφερθώ στα θέματα που θεωρώ πιο σημαντικά και στις εξουσίες βεβαίως του Κοινοβουλίου. Ασφαλώς δεν πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισμός όπως αναφέρθηκε. Συμφωνώ απολύτως στον πολιτικό συντονισμό, στην ε, λήψη υπόψη διαφορετικών παραδόσεων νοοτροπιών στα θέματα της διπλωματίας που ανέφερε ο κύριος Λάμπστορφ, ο κύριος Χόποντα επίσης το ρόλο των αναπληρωτών της κυρία Άστον και των επιτρόπων. Θα ήθελα να δω εδώ τι έχετε να μα πείτε συγκεκριμένε προτάσεις. Πάντως να μην δοθεί εντύπωση ότι ο Επίτροπος είναι αναπληρωτής του αναπληρωτή της είπα τη εκπροσώπου. Άλλο ότι έχουμε να κάνουμε μάλλον μια πολιτική εκπροσώπηση. Ούτε ότι χάνει κάποια από τις αρμοδιότητες ή τις προνομίες της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω λοιπόν ότι ίσως με πιο καλή διατύπωση το κείμενο θα ήταν δυνατόν να ε, επιληθούν κάποιες ε, παρεξηγήσεις. Θα το δω με τον κύριο Φερχόφστατ. Πάντως θα ήθελα να πω ότι μπορέσαμε μέχρι τώρα να συνεργαστούμε πολύ καλά, να διατηρήσουμε ένα καλό επεδό ε, συμφωνίας και συνένεσης, πράγμα το οποίο ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και στις ε, στη φάση των τροπολογιών, όχι μόνο από τι διάφορε επιτροπέ που θα εμπλακούν στην τι αλλά και σε ολόκληρο το επίπεδο του Κοινοβουλίου, ώστε να έχουμε όσο δυνατόν τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη για το κείμενο αυτό, για την έκθεση όταν είναι έτοιμη. Επίσης, ε, είπατε, είπε μια στάλφο ότι θα πρέπει να έχουμε και προσωπικό από την Υπουργεία Αναπτύξεω. Ναι. Βεβαίω και φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει δεκτό με πολύ ενθουσιασμό και από αρκετές ε, πρωτεύουσες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι παράξενο βέβαια το ότι κάποιοι ε, οι πολλοί άριθμοι, μάλλον με μερικέ χιλιάδε υπάλληλοι έρχονται εδώ για να παίρνουν του υψηλού ευρωπαϊκού μισθού, αλλά στη συνέχεια δεν υποστηρίζουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα γιατί θεωρούν ότι δεν είναι αυτή η δουλειά του. για τις απαντήσεις ή για τις αποφάσεις. Αποφάσεις λαμβάνονται στο επίπεδο που πρέπει να ληφθούν. πίνα. Αναπτυξιακή Επιτροπή, Επιτροπή. Η ύπατη αρμοστία, η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων με τον, ανα... για το, με τον Επίτροπο των Αναρμόδιων για την Ανάπτυξη λαμβάνει τι αποφάσει για, για τα θέματα τη ανάπτυξη. Όχι μόνο στο Επίτροπο, όχι μόνο τη ύπατη εκπρόσωπο, σε συνεργασία. Συλλογικά λαμβάνονται αυτέ οι αποφάσει για την αναπτυξιακή πολιτική. Ούτε μπορεί όμω μόνη τη, είπατε, εκπρόσωπο να κάνει μόνη τη προτάσει για την αναπτυξιακή πολιτική, πάντα σε συνεργασία με τον αρμόδιο για την ανάπτυξη επίτροπο. Συλλογικά αποφασίζει η Επιτροπή και σε περίπτωση σύγκρουση το συλλογικό όργανο. Όχι μεμονωμένο κάποιο, πάντω όχι είπατε εκπρόσωπο μόνη τη. η πραγματογνωμοσύνη στην οποία αναφέρθηκε άλλο συνάδελφο. Την γνωρίζω πάρα πολύ καλά, την έχω διαβάσει, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι σωστή. Είναι σφαλμένη βάση της. πρέπει να έχουμε συνέπεια ως προς την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα συνέπεια και συνοχή με την εξωτερική δράση, με την εξωτερική πολιτική. Και γι' αυτό προβλέπετε και για τη σχετική υπηρεσία, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, ότι θα υπάρχουν και οι ε, υπάλληλοι της Επιτροπής. Κατά πλειονότητα θα είναι υπάλληλοι της Επιτροπής το προσωπικό που θα επανδρώσει αυτήν την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Στόχο μα είναι να μπορέσει να γίνει δουλειά σωστά. Είπατε και εσείς ότι έχουμε να κάνουμε διαφορετικές νοοτροπίες και παραδόσεις. Πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε ώστε να έχουμε μια ε, πολιτική συνεκτική. Την τελική απόφαση θα τη λαμβάνει ή το Συμβούλιο ή η Επιτροπή Συλλογικών Οργανών με την περίπτωση. Για τον κύριο Σαλαφράγκα ναι, το πολιτικό, το πολιτικό κοινοβούλιο πολιτικά αποφασίζει, πολιτικά ε, δρά. Δεν έχει εκτελεστικό ρόλο το κοινοβούλιο, ρόλο νομοθετικό έχει, ρόλο ελέγχου έχει, ρόλο δημοσιονομικό έχει, αποφασίζει το προπολογισμό και, όπως είπα, πολιτικό πάνω απ' όλα, τίποτε άλλο δεν έχει. Βέβαια, ε, όπω είπα και πριν, το να επιδιώκουμε κάποιου στόχου έχει νόημα. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει διαβούλευση, επαφή με, με, το Κοινοβούλιο και το συντονισμό σε πρόωρο στάδιο, έτσι ώστε να έρθει η ώρα το Κοινοβούλιο με τον προπολογισμό, παραδείγματι, να δώσει το πράσινο φω για τα θέματα του προσωπικού, για τα, κονδύλια δηλαδή για το προσωπικό. Θα πρέπει να είναι εγκαίρω ενήμερο ώστε να μπορεί να παρακολουθεί αυτή την υπόθεση ώστε να δώσει το πράσινο φως. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει ο έγκαιρος συντονισμός. Αυτό είναι ο στόχο που επιδιώκουμε τουλάχιστον εμεί. Με τις διαβουλεύσει, με την έγκαιρη ενημέρωση, να είναι δυνατόν το κοινοβούλιο να εκφράζει τι θέσει του έγκαιρος ώστε να μην υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις στο τέλος. Διότι στο τέλος μπορεί η έκπληξη να είναι πάντοτε η αρνητική απάντηση. Πρέπει να σας πω ότι βρίσκω εξαιρετικά χρήσιμο αυτό το ε, παιδαγωγικό μέσον της διαδικασίας συναπόφασης, γιατί βοηθάει πολύ ορισμένους να μαθαίνουν να συνεργάζονται. Επίσης για το sui generis. Τι σημαίνει sui generis. Στην ε, διάσκεψη για τη συνταγματική συνθήκη, όσο να θυμάστε, είχαμε συζητήσει διάφορα θέματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε πει, είχε συζητηθεί το θέμα του sui χαρακτηριστικό. Ε, sui ωστόσο δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεται από τον έλεγχο, ότι βγαίνει εκτός κάποιου συγκεκριμένου θεσμικού κύκλου. Δηλαδή, ο ναι, είναι ένα σουιγγένερισόν όργανο, υπάγεται όμω πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σουιγγένερη είναι η υπηρεσία εξωτερική δράσεω, ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απολύτω ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη αρχή. Είναι ένα όργανο εξωτερική πολιτική μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να χαρακτηριστεί κάποια υπηρεσία σου generis, απαιτείται να υπάρχουν και σοβαροί λόγοι γι' αυτό. Σοβαροί λόγοι είναι ότι έχει ένα διαφορετικό από τα συνηθισμένα, από τα ιωθώτα χαρακτήρα. Έχει κάποια στοιχεία που τη διαφοροποιούν από το, από το μέσο όρο. Εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπω πουθενά εγώ μέχρι τώρα, ούτε από την κυρία Άστον, ούτε από το Συμβούλιο, πρόταση που να δίνει ερμηνεία του sui generis διαφορετική από αυτήν την οποία εννοώ εγώ, δηλαδή την υπαγωγή πάντως στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν έχει ο κ. Χριστόφος μια διαφορετική γνώμη, τι να πω. Αν θέλει ίσως να το σημείο 6 και στα θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό. Νομίζω ότι και εκεί θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς ότι μπορεί να γίνει μέσα στον κοινό μας προϋπολογισμό στον απλό, στο, στο δεδομένο μα προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. ένα ειδικό τμήμα, αφού είναι σου generis η υπηρεσία. Ένα ειδικό τμήμα, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βγει έξω από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ θα τα πούμε αυτά τα πράγματα, πώ θα ισχυριστούμε κάτι τέτοιο. Πώ θα διαπραγματευθώ μετά για το, για το Συμβούλιο. Νομίζω ότι πρέπει ο καθένα να είναι σε θέση να διαπραγματευτεί τι τις θέσεις χωρίς να αποκλείει καμία δυνατότητα μετακίνησης. Ευχαριστούμε. Ε, ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Φερχόφστατ ζήτησε να παρέμβει. Σας παρακαλώ να είσαστε ιδιαίτερα σύντομος. Ευχαριστώ. Απλώς θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που είπε ο κύριος Βρόκ για το δημοσιονομικό σκέλος για το θέμα τμήμα 3, τμήμα 6. Δεν είναι σωστό ότι υπονομεύουμε τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν η υπηρεσία υπο, υπαχθεί στο τμήμα 3. Λάθος. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη διαπραγμάτευση γιατί αυτόματα κατοχυρώνονται. Και μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια συντάσσοντας ένα ξεχωριστό κεφάλαιο του τμήματος 3 με τις διαφορετικές δυνατότητες. Θα μιλήσουμε για το κεφάλαιο 13, 23β, 26. Υπάρχουν πολλές και διάφορες δυνατότητες γι' αυτό. Και το πλεονέκτημα όλων αυτών είναι ότι παραμένει στο κοινοτικό τμήμα του γενικού προϋπολογισμού. Και δεν είναι και άνευ προηγουμένο, γιατί η ΚΕΠ αυτή τη στιγμή που εντάσσεται στο τμήμα 3. Δεν υπάρχει ξεχωριστό τμήμα για την ΚΕΠΑ. Και η ΚΕΠΑ είναι νομίζω ότι το, είναι το επιχείρημα που μπορούμε να παρουσιάσουμε στο Συμβούλιο και το παράδειγμα για να αποδείξουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να υπαχθεί στο τμήμα 3. Τι φοβόμαστε θέλουμε να κάνουμε ξεχωριστή υπηρεσία στον προϋπο... Ε, ξεχωριστό τμήμα στον προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα δημιουργήσουμε ένα τεράστιο προηγούμενο για το μέλλον. Γιατί κάθε φορά που θα ιδρύουμε μια υπηρεσία, ή έναν οργανισμό, λέμε Α, και η ΕΔ είναι ξεχωριστή, το ίδιο πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Θέλουμε δύο νέου οργανισμού για την ε, χρηματοπιστωτική εποπτεία και οι τρεις οργανισμοί θα χρηματοδοτηθούν εν μέρη από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και εν μέρη από τα κράτη-μέλη. 60% του προϋπολογισμού των οργανισμών θα χρηματοδοτηθεί από τα κράτη-μέλη. Ποια θα είναι η αντίδραση αν κάθε φορά προβλέπουμε ξεχωριστό τμήμα όταν το Συμβούλιο ή τα κράτη-μέλη θα έχουν το λόγο τους ε, στους οργανισμούς αυτούς. Θα πούμε, α, έχουμε το παράδειγμα της ΑΕΕΒ και για αυτές τους οργανισμούς θα πρέπει να εκπέσουν από το τμήμα 3 και να μπουν σε ξεχωριστό τμήμα. Αν ξεφύγει η ΕΙΕΔ από το τμήμα 3 και ενταχθεί σε ξεχωριστό τμήμα, θα δημιουργηθεί προηγούμενο και θα, το, θα επικαλείται το Συμβούλιο αυτό το επιχείρημα, ώστε κάθε νέος οργανισμός να υπάγεται σε ξεχωριστό τμήμα. Στο μέλλον μπορεί να έχουμε και οργανισμό ενέργειας. Και πάλι θα μας πει από τη στιγμή που ενέχεται το Συμβούλιο και πάλι θέλουμε ξεχωριστό τμήμα. Οπότε θα εκενώσουμε με τον τρόπο αυτό περιεχομένου την κοινοτική μέθοδο. Βγάζοντας πολιτικές από το τμήμα 3. Αυτό είναι ο φόβος μας, περί αυτού πρόκειται. Και, το, και, το, και στην ΚΕΠΑ ενέχεται το Συμβούλιο, αλλά παρόλα αυτά η ΚΕΠΑ εντάσσεται στο τμήμα 3. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Σας ευχαριστώ όλοι γιατί ε, συνεισφέρατε έμπρακτα και ουσιαστικά στη συζήτηση. Το επόμενο θέμα είναι η πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Πρόκειται η δεύτερη συζήτηση επί του σχεδίου ψηφίσματος. Προηγουμένως η Επιτροπή είχε συζητήσει θέματα που είχε θίξει η συγγήτρια, η κυρία Πάκα, και η σημερινή συζήτηση σχετίζεται με την ε, τροπολογία 194 στην ε, έκθεση της εισηγήτρια. Σας παρακαλώ λίγη ησυχία για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Υπό το φως των συζητήσεων η εισηγήτρια θα συζητήσει με τους σκιώδεις για να συμφωνήσουν σε τροπολογία συμβασμού. Το λόγο έχει η κυρία Πάκ. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Äh, Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επιμείνουμε επιμακρών στην έκθεση αυτή, γιατί ήδη είχαμε διεξοδική συζήτηση. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι κατέθεσαν τροπολογίες, ε, συνολικά 194 στον αριθμό. Βλέπετε ότι είναι πληθώρα οι τροπολογίες, δεν θα είναι εύκολο να συμφωνήσουμε, ούτε μπορώ να τις δεχτώ όλες. Προσπάθησα να καταρτήσω κάποιες συμβαστικές τροπολογίες και κατά την εβδομάδα του Στρασβούργου θα προσπαθήσω να τις παρουσιάσω στους συναδέλφους προκειμένου να εξοικειωθούν με αυτές. Έλαβα κάποιες τροπολογίες που βελτιώνουν την έκθεση ή την εμπλουτίζουμε κάποια σημεία που δεν είχαν περιληφθεί αρκετά. Παρακαλώ λίγη ησυχία στην αίθουσα για να μπορέσω να συγκεντρωθώ. Κύριε Βερχόφστατ, δεν είναι πολύ ευγενικό απέναντι στην εισηγητριά μας να δημιουργούμε τέτοια φασαρία στην αίθουσα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Καινοτομίε είναι τα θέματα των μέσων μαζική ενημέρωση, το θέμα των μειονοτήτων, που επισημαίνεται και ενισχύεται χάρη σε ορισμένε τροπολογίε, το θέμα τη δικαιοσύνη. Επίση ενισχύεται, η πάταξη τη διαφθορά. Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία δεν είναι επίμαχα, και μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτά σε ικανοποιητικέ συμβαστικέ τροπολογίε. Βέβαια, κάποιε τροπολογίε ε, ζητούν διαγραφή διαφόρων παραγράφων και είναι απαράδεκτε, κατά τη γνώμη μου. Βέβαια, θα το κρίνει η πλειοψηφία τελικά, θα εγκριθούν ή όχι. Θα γίνουν και κάποιες αλλαγές. Θα υποβληθούν και προφορικές τροπολογίες στα πλαίσια των συμβαστικών μας τροπολογιών. Για παράδειγμα, κάποιες χώρες ε, που δεν έχουν ε, αναγνωρίσει ακόμη την ανεξαρτησία θα πρέπει να προσέξουμε όταν επισημαίνω αυτές τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών που έχουν εγκρίνει και των άλλων που δεν έχουν εγκρίνει. Επίσης, το θέμα των μειονοτήτων θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης μεταχείρισης. το να αναφέρουμε ονομαστικά τις μειονότητες δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο. Προτιμώ να μιλούμε γενικά και όριστα για τις μειονότητες, για την εσφαλμένη αντιμετώπιση, μεταχείριση των μειονοτήτων ή διακριτική μεταχείριση βάρος μειονοτήτων. Αλλά γενικά, παρακαλώ σταματήστε τις ε, συνομιλίες, τις ιδιωτικές, γιατί δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, λέει η συγκεντρία. Σε διάφορα σημεία της έκθεσης βέβαια. Κατονομάζω συγκεκριμένα, συγκεκριμένους. Καλύτερα να μιλούμε γενικά για τους θεσμούς, να μιλούμε για τον Πρωθυπουργό ή για άλλους θεσμούς, αλλά να μην αναφέρουμε ονομαστικά τέτοιους εκπροσώπους. Καλύτερα είναι πιο ουδέτερο το κείμενο. Γιατί πολλές τροπολογίες ε, αναφέρουν αυτές τις προσωπικότητες, συγκεκριμένα ονόματα προτιμώ να είμαστε πιο αμερόληπτοι και ουδέτεροι, να μιλούμε περισσότερο για θεσμούς παρά για ονόματα, για συγκεκριμένες προσωπικότητες. Θα προσπαθήσω στις συμβαστικές μου τροπολογίες να συγκεράσω πολλές από τις ε, τροπολογίες αυτές και πριν ξανασυζητήσουμε το θέμα στο Στρασβούργο θα συναντήσω και τους κοιόδης συγητές. Υπάρχει και το θέμα του είπατε εκπροσώπου. Προτιμώ να είμαστε πιο συνετοί, αποφασιστικοί μεν αλλά συνετοί, αποφασισμένοι αλλά συνετοί. Θα το δούμε και αυτό. Για τη Σρεμπρένιτσα, δεν την αναφέρω καν στην έκθεσή μου. Πολλοί σκιώδεις συγητές επέμειναν να τη συμπεριλάβω να αφιερώσω κάποιους παραγράφους στη Σρεμπρένιτσα και ομολογώ ότι έχουν δίκιο. Δεν αρκεί μόνο να μιλούμε για τη Σερβία. Θα πρέπει να ενταχθούμε στο συγκεκριμένο πλαίσιο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω αυτό το θέμα σε μια συμβαστική τροπολογία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη Βοσνία Ζεγοβίνη καταρτίζοντας τόσες πολλές τροπολογίες. Το θέμα της απελευθέρωσης, κατάργησης των θεωρήσεων αναφέρθηκε από πολλούς συναδέλφους και θα φροντίσω να βρω μια ικανοποιητική διατύπωση που θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, χωρίς να γύρω όμως ελπίδες ή προσδοκίες που θα είναι φρούδες για τον πληθυσμό. Πρέπει να, δω, να προσπαθήσουμε να βρούμε μια μέση οδό και τίποτε άλλο. Επίσης έχουμε το ζήτημα του λαθρεμπορίου, το, της εμπορίας ανθρώπων. Ε, είναι ένα ιδιάζων υποτίθεται κράτος ε, στην υπόθεση αυτή η Βοσνία γιατί είναι και κράτος διελεύσεως και κράτος προελεύσεως. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς διατυπώνουμε αυτούς τους όρους ώστε να μην ε, έχουμε ε, ανεπιθύματα αποτελέσματα ή εντυπώσεις. Και θα ήθελα επίσης να σημειώνω ότι η Βοσνία καλείται τώρα να ε, προχωρήσει στην ένταξη, στο πρόγραμμα μάλλον ένταξης ε, του ΝΑΤΟ διάφορα στοιχεία τα οποία θα μας απασχολήσουν ασφαλώς προσεχείς δύο-τρεις εβδομάδες. Σας ευχαριστώ θερμά και περιμένω από τους συναδέλφους να ακούσω εάν συμφωνούν τουλάχιστον ως προς τη διαδικασία και ίσως μπορούμε να βρούμε και συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε το λόγο στους Σκιώδης τώρα. Η κυρία Σαρτζεντίν είναι η, η πρώτη ομιλήτρια. For, for this, um, for this explanation. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις επεξηγήσεις. Ευχαριστώ κυρία Πακ Συμφωνώ ότι το ψήφισμα της Βοσνίας είναι πολύ καλό και βελτιώνει την ανάγκη ύπαρξης ανεξάρτητων ε, μέσων γιατί οι... εμείς οι πράσινοι προσδίδουμε μεγάλη σημασία στη δημοκρατία. Δεν θα ήθελα να φέρθω σε ονόματα γιατί μιλάμε. Μιλάμε για ανθρώπους που φέρουν ονόματα πρέπει να καταφέρθουμε κατά των διακρίσεων ευάλωτων ομάδων στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Εμείς υποβάλαμε τροπολογίες σε σχέση με την προστασία ε, ομοφιλοφίλων και όλων αυτών των κατηγοριών τη στιγμή που δεν μιλάμε για μεγάλες εθνοδικές ομάδες. Εάν θέλουμε να έχουμε μια καλή διαδικασία ένταξης της ε, Βοσνίας, τότε θα πρέπει να είμαστε σαφείς για το τι μιλάμε και ε, ως προς την καταπολέμηση των διακρίσεων και στο, στα εθνοτικά και στις ε, σεξουαλικές προτιμήσεις στην Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών, όπου μιλήσαμε για την απελευθέρωση των θεωρήσεων στη Βοσνία, είδαμε ότι υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις, αλλά πιστεύω ότι η Βοσνία Ερζεγοβίνη θα μπορέσει να καλύψει τα κενά στις, ε, στα πλαίσια αυτών των διαδικασιών για την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων μετά το καλοκαίρι. Ε, λυπάμαι γι' αυτό, αλλά θα γίνει μετά το καλοκαίρι. Άρα οι Βόσνοι θα μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για την σταθεροποίηση της περιοχής. Ευχαριστώ την κυρία Πακ και αναμένω τη συζητήση μας την επόμενη εβδομάδα για να δώσουμε τελική μορφή στο ψήφισμα. Η κυρία Μπόσκουρτ από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία ΠΑΚ για τα εισαγωγικά της σχόλια σε σχέση με τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στην έκθεση και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προσβλέψουμε σε μια πολύ καλή έκβαση. Πολλά θα πρέπει να προστεθούν στην έκθεση έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα από πλευρά σοσιαλιστών έχουμε υποβάλει μια σειρά ε, τροπολογιών όπως για την ε, οικονομική ολοκλήρωση, απασχόληση και κοινωνική ένταξη. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία όταν μιλάμε για τη διαδικασία ολοκλήρωσης και συμμετοχής των διαφόρων εθνοτικών ομάδων στη Βοσνία. Γιατί όλα ξεκίνησαν από την οικονομική συνεργασία και βεβαίως θα πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές ως προς τις μειονότητες. Έχω μία ερώτηση και ελπίζω να απαντήσετε, διότι είπατε ότι όλες οι μειονότητες θα πρέπει να αναφέρονται ως μία ομάδα και να μην τις κατονομάσουμε χωριστά. Αν λάβουμε υπόψη όμως τους Ρωμά που αναφέρονται ρητά σε τροπολογίες, τότε έχουμε να κάνουμε με μία ειδική κατηγορία που αντιμετωπίζει ειδικά προβλήματα, που έχει ένα ευρωπαϊκό εύρος. Άρα όταν μιλάμε για μία μεγάλη εθνοτική ομάδα, τότε χάνουμε από το οπτικό μας πεδίο τους Ρωμά, για παράδειγμα. Ως προς το Σύνταγμα της Βοσνίας, έχουν υποβληθεί τροπολογίες και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είπε ότι δυστυχώς το Σύνταγμα οδηγεί σε πολλαπλές διακρίσεις ως ε, έχει. Όπως έχει διατυπωθεί επίσης, ε, μιλήσατε του, για αυτούς που απομονώνονται στο εσωτερικό της χώρας. Πολλοί βεβαίως δεν μπορούν να επιστρέψουν στις αιστείες τους, είναι ε, δηλαδή απομακρυσμένοι Ως προς το θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων, ελπίζουμε να καταφέρουμε κάτι πριν από τις εκλογές τον Οκτώβριο. Ε, παρενέβησαν οι σκιώδεις. Τώρα θα παρέμβουν οι συνάδελφοι Ήμπραζης, ε, Αγκουράκης, και Τάλεκ. Ήμπραζιτς. Tackar ordförande. Ehm, jag ska försöka fatta mig väldigt kort. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι λακωνικότατη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ντόρις για την ε, πολύ καλή της ε, έκθεση. Υπάρχουν πολλά σημεία που επαναθεωρήσαμε και συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να αναζητήσει συμβαστικέ λύσει για τα νομικά ζητήματα, για τα θέματα των μειονοτήτων, για την ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση, για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, για θέματα που μα βρίσκουν σύμφωνου. Εκεί μπορούμε να καταλήξουμε στη συμβαστική συμφωνία, συγκερνώντα τι άλλε τροπολογίε. Και συμφωνώ με το αρχικό κείμενο τη ε, Ντόρι σε πολλά θέματα. Θα πρέπει να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Προτιμώ την αρχική διατύπωση της δόρης για πολλά σημεία και δεν θα πρέπει να ενδώσουμε και να υποκύψουμε στις πιέσεις. Και σε προηγούμενα ψηφίσματα είχαμε πει πολλά για τη Βοσνία Ριζεγοβίνη, το κείμενό μας ήταν σαφές και είναι καλό να είμαστε και επικριτικοί μερικές φορές. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς με αυτά που λέμε. Θα πρέπει να ορθώσουμε το παράστημά μας και να έχουμε το θάρρος της γνώμης μας, ακόμη και της επικριτικής, όταν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι η Ντόρις θα πρέπει να δείξει αποφασιστικότητα, να εμείνει στην αρχική της θέση σε πολλά σημεία και να μην αλλοιωθεί το ψηφισμά της. Γιατί αν είμαστε υπερβολικά διπλωματικοί και ρίχνουμε νερό στο κρασί μας, δεν θα είμαστε αποτελεσματικοί. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να διατρανώσουμε τη γνώμη μας, γιατί πλησιάζουν και οι εκλογές στη Βοσνία και όπου υπάρχει δυσαρέσκεια και δυσφορία θα πρέπει να την ε, εκφράσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αγκουράκης, εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, η ομάδα μας θα καταψηφίσει φυσικά αυτή την έκθεση παρά τις τροπολογίες που έχουν γίνει. Ε, για τον πολύ απλό λόγο ότι και οι τροπολογίες δεν αντιμετωπίζουν το βασικό πρόβλημα της χώρας αυτής που είναι η νεοαπικιοκρατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία πολιτική δεν επιτρέπει στη Βοσνία Τζεγκοβίνη, στο λαό της Βοσνίας Τζεγκοβίνης να γίνει κυρίαρχος της χώρας του. Έχουμε τη γνώμη ότι θα έπρεπε το Ευρωκοινοβούλιο να ζητήσει να τεθεί ένα τέρμα στην στρατιωτική παρουσία, στρατιωτική κατοχή θα έλεγα εγώ της ε, ε, Βοσνίας Ατζεγκοβίνης, όπως επίσης θα έπρεπε το Ευρωκοινοβούλιο να ζητήσει να κλείσει εδώ και τώρα το γραφείο του ΙΠΑ, του αρμοστή του, των Ηνωμένων Εθνών και το γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία Τζεγκοβίνη. Κύριε Πρόεδρε, ε, όσο καιρό δεν αντιμετωπίζεται στη ρίζα του το πρόβλημα της χώρας αυτής, τα πολλά προβλήματα στα οποία αναφέρθηκε η κυρία Ντόρις Πακ και υπάρχουν στη χώρα αυτή, θα διαιωνίζονται, θα γίνονται ακόμα πιο οξυμένα και θα το δείτε, σε μερικά χρόνια θα είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση, διότι κακά τα ψέματα. Δεν λύνεται το πρόβλημα της Βοσνίας Ετζεγκοβίνης με το να απελευθερωθούν οι βίζες και να, μπορούν, ε, να μπορεί ο πληθυσμό της χώρας αυτής να κυκλοφορεί ελεύθερα. Στην ουσία η εισηγήτρια μας λέει ότι δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα της χώρας, γι' αυτό το λόγο ας πάνε οι Βόσνοι ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να βρουν μια καλύτερη ζωή. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή την προσέγγιση, γι' αυτό και νομίζουμε ότι τα βασικά ζητήματα έχουν να κάνουν με το να κλείσουν αυτές οι υπηρεσίες και να δοθεί δυνατότητα στους Βόζιους να καθορίσουν μόνοι τους την τύχη τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τη συνάδελφο Ντόρι Σπακ για την ε, πολύ σωστή έκθεσή της που χαρακτηρίζεται από υψηλό επαγγελματισμό και αντικατοπτρίζει την ε, μακρόχρονη ενασχόληση και αφοσίωση της Doris Πακ στη χώρα αυτή. Μερικές φορές ακούμε ότι η Βοσνία Ζεγοβίνη είναι πλήρως λειτουργών κράτος και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας έχει συμπεριληφθεί η Βοσνία Ζεγοβίνη στη συζήτηση για την ε, λήψη αποφάσεων πολλών σημαντικών θεμάτων. Και από τη στάση του Συμβούλιο Ασφαλείας φαίνεται ότι η Βοσνία Ζεγοβίνη είναι ένα κράτος που λειτουργεί εύρυθμα. Όπως λοιπόν λειτουργεί προς τα έξω, καλό θα ήταν το ίδιο εύρυθμα να λειτουργεί και εσωτερικά. Και η εικόνα που δίνει στον έξω κόσμο να έχει μία αντανάκλαση στην εσωτερική πραγματικότητα της Βοσνίας. Η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ θα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα και θα δημιουργήσει Ευκαιρίε πρόοδου και μετά τις εκλογές. Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο όμως αυτή τη στιγμή είναι η ρητορική που ακούμε αυτή τη στιγμή εντός της Βοσνίας σε Πριν από λίγε μέρες ε, συγκλονίστηκα ακούγοντας ε, ζωντανές δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Ρεπούμπλικα Σέρψτα στο Ζάγκρεπ σε έναν ε, αγώνα μπάσκετ που μάλιστα επισκέφθηκε ανεπίσημα Παρακολούθησαν επίσημα και όταν ρωτήθηκε ποιον θα υποστηρίξει αν στον τελικό η Βοσνία Ζεγοβίνη είναι αντιμέτωπη με την Κροατία. Και είπε ανενδίαστα ότι θα υποστήριζε την Κροατία γιατί δεν είναι ένθερμος οπαδός της Βοσνίας ζεγοβίνης. Δεν ξέρω ούτε μία χώρα της Ευρώπης όπου εκπρόσωπος της, είπα, εκπρόσωπος εκτελεστικής εξουσίας οποιασδήποτε χώρας θα έκανε τέτοια δήλωση ότι θα προτιμούσε να υποστηρίξει μια άλλη χώρα και παρόλα αυτά να παραμείνει στη θέση του. Αυτό πραγματικά είναι ανάξιο και της πολιτικής, του πολιτικού βίου, αλλά και της κυβέρνησης. Δεν μπορεί κάποιο που περιφρονεί την πατρίδα του να εξακολουθεί να παραμένει σε ένα τέτοιο υπατό αξίωμα. Νομίζω ότι είναι προσβολή όχι μόνο κατά της Βοσνίας, αλλά και κατά των ε, πολιτιστικών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοια προβοκάτσια, τέτοια προκλητική συμπεριφορά δημιουργεί πολύ αρνητικές συνέπειες και θα πρέπει να συλλητευθεί και να καταδικαστεί στην Βοσνία. Πολλό δε μάλλον που έχουμε και προεκλογική εποχή. Σε ό,τι αφορά τη ρητορική για τα, για τα θύματα των Βαλκανικών πολέμων στη Βοσνία Ριζγοβίνη, αυτή η ρητορική χρησιμοποιείται μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Έχουν ε, κατασκευαστεί νέα μνημεία και αποτείεται φόρος τιμή σε νέα θύματα, αλλά μόνο και μόνο για ψηφοθυρικούς λόγους. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στη συνδιάσκεψη του Σαράγεβα που θα γίνει στις 2 Ιουνίου. Και αν υπάρχει δυνατότητα να συμφωνήσει η Βοσνία και να προσεγγίσει περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματικά θα ήταν μια αξιέπαινη προσπάθεια και χρήζει υποστήριξης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφη κυρία Πακ και να τη συγχαρώ για τη δουλειά της, όπως και οι συνάδελφοι. Είναι σαφές ότι ε, είναι έμπειρη στα θέματα ιδιαίτερως της ε, πρώην Γιουγκοσλαβίας, της Βοσνίας Τρισεκοβίνης ιδιαίτερως Βλέπω με χαρά λοιπόν ότι θα υποφαληθεί το Κοινοβούλιο από την εμπειρία αυτή. Και δεύτερον, έχουμε σήμερα την 30η επέτειο του θανάτου του στρατάρχη Τίτο και ορισμένοι από εμάς θυμόμαστε ακόμα την εποχή ότι λειτουργούσε το κράτος αυτό της Ιουγκοσλαβίας όσο ήταν ζωντανός και όσο το καθοδηγούσε ο Τίτο. Και χρειάστηκαν μόλις 10 χρόνια για να διαλυθεί το κράτος από το θάνατό του. 10 χρόνια από το θάνατό του για να διαλυθεί το κράτος. Εδώ ακριβώς ξεκινούν και τα προβλήματα και τα δεινά της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Εδώ ακριβώς εντοπίζονται και οι δικές μας ευθύνες δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν ε, πώς είναι δυνατόν οι συναδέλφοι από την άκρα αριστερά να πιστεύουν ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε στη μοίρα της τη Βοσνία, να την αφήσουμε να διαλυθεί τελείως. Διότι θα πρέπει να διερωτηθούμε πρώτα απ' όλα εάν είναι σε θέση να παρακολουθήσει την, ε, τις εξελίξεις η Βοσνία, αν έχει αρκετά, ε, αρκετό δυναμικό, αρκετές δυνατότητες η Βοσνία για να προχωρήσει προς ένα νέο δρόμο ανοχής και αλληλοκατανόησης. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις ακόμη σε επίπεδο Βοσνίας και γι' αυτό θα πρέπει να την υποστηρίξουμε, να τη στηρίξουμε με κάθε, κάθε μέσο. Είναι ξέρετε το ψήφισμα λοιπόν, όπως είπα και νωρίτερα, διότι ασχολείται με θέματα ουσίας, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη διαφθορά, τις μειονότητες και άλλα θέματα. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω άλλο ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική πτυχή, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα καθεστώς θεωρήσεων, ειδικά για τη Βοσνία, ώστε να εκπαιδεύσουμε τους νέους της Βοσνίας ε, να προχωρήσουν για το μέλλον, προς το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τάλας. Ο κύριος Μίρελ, που είναι ε, διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση. Ε, ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα θέλαμε και εμείς να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε στο βαθμό του δυνατού, ίσως και να εμπλουτίνουμε αυτή την εξαιρετική έκθεση με τις παρατηρήσεις μας, δύο τον αριθμό. Η μία αφορά το Σύνταγμα της ε, Βοσνίας Ερσεγοβίνης, το οποίο παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και την Συμφωνία Εμπορίου, την SAA, στο άρθρο 2 και νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να επισημανθεί και αυτό μέσα στο κείμενο. Και δεύτερη παρατήρηση. Καθεστώς ε, θεώρηση, απελευθέρωση τους ε, θεώρησης. αφού δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη τα ορόσημα, παραμένουν ορισμένα, θα ήταν ε, καλό να δοθεί, μια, να δοθεί σαφής υποστήριξη προς τις αρχές στον στόχο αυτών, ώστε να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους. Η κυρία Πάκ να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο. Για την κυρία Μποσκούρτ θα ήθελα να πω ότι βεβαίως είναι πολύ σημαντική η δουλειά και η ανάπτυξη σχεδίων, αλλά χρειάζεται και μια εσωτερική αγορά μέσα στη Ποσνία. Στη Βοσνία Ερσεγοβίνη δεν υπάρχει εσωτερική αγορά, εάν το πιστεύετε εάν το πιστεύετε. Κάτι που θα μπορούσε να εξασφαλίσει νέε θέσει Κάτι που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κάνουμε πρώτα απ' όλα. Και βεβαίω στι δικέ μου τροπολογίε, μάλλον θα έλεγα σε αυτό που έχω υπόψη για, την, για τις συμβαστικές τροπολογίες, Έχω και τους ε, Ρωμά, τους Τσιγκάνους υπόψη, αλλά και μειονότητες είναι και άλλες. Και κυρία Μποσκούρτ, οι γυναίκες δεν είναι μειονότητα, το μισό της, ε, των κατοίκων είναι. Έτσι λοιπόν όταν μιλούμε για μειονότητες, τα ασεξουαλικά, η γενετήσια προβλήματα, η γενετήσια συμπεριφορά, ε, να μας λέτε ότι θα πρέπει να γίνονται ανεκτά κτλ, αν θα πρέπει να τα απαριθμίσουμε, ίσως πρέπει να το δούμε λίγο αργότερα όλα αυτά. Επίσης, το Σύνταγμα το αναφέρω ξεκάθαρα, αλλά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά αυτό που είπε ο κ. Σαμιρέλ τώρα για το δικαστήριο, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την υπόθεση σχετική με το εξωτερικό εμπόριο, ναι, έχουμε προβλήματα τα οποία πρέπει να υπογραμμίσουμε ε, και θα έπρεπε ουσιαστικά να έχουν προχωρήσει πριν από τις εκλογές, δυστυχώς όμως πια μένει χρόνος για, μέχρι τις εκλογές για να αντιμετωπιστούν αυτά. Και κύριε Μιρέλ. Έχουμε φτάσει στο Μάιο. Ιούνιο για να περάσει την Ολομέλεια και μα μένουν τρει μήνε μέχρι τι εκλογέ. Λέτε να, προβάλλουμε, να προλάβουμε. Επιθυμίε μπορούμε να εκφράσουμε φυσικά, αλλά μάλλον δεν μπορούμε να επηρεάσουμε πια την κατάσταση. Δυστυχώ, δυστυχώ αφήσατε πολύ χρόνο να πάει χαμένο. Έτσι είναι τα πράγματα. Για το συνέλφα από του κομμουνιστέ. Θα ήθελα να πω ότι οι προτάσεις, οι ιδέε για προσφορία αρρωγή στο κράτο αυτό νομίζω ότι είναι επονίδιστες δεν ε, θα έπρεπε να μιλούμε όχι για Ελλάδα ούτε για τίποτα με αυτά που μας προτείνεται να δώσουμε στη χώρα αυτή ως βοήθεια. Δηλαδή να τους αφήσουμε να καταποντιστούν, ναι. Εμείς προσπαθούμε να τους στηρίξουμε και προς την ορθή κατεύθυνση. Και αυτό που, κάνουν εκεί, αυτό που κάνουμε εμείς στη Βοσνία είναι να τους βοηθήσουμε να σταθούν στα πόδια τους πρώτα απ' όλα. Αυτά έχω προτείνει μέσα στην έκθεσή μου. Αυτό που δεν έχω προτείνει μέσα στην έκθεσή μου είναι ότι η, η απλή και μόνη κατάργηση της υποχρέωσης για θεώρηση διαβατηρίου δεν θα σώσει τα πράγματα. Αυτό δεν το λέω. Όχι. Δεν θεωρώ ότι πρόκειται να του σώσει. Α δούμε πώ θα ήταν τα πράγματα αν υπήρχε δυνατότητα να ταξιδεύουν βεβαίω. Α δούμε ότι υπάρχει στη Βοσνία Ερσεγοβίνη εκπροσώπηση τριών διαφορετικών εθνοτήτων Και πώς μπορούμε να πούμε για τις δύο από αυτές τις εθνότητες, γιατί σε τελευταία ανάλυση ούτε η Κροατία είχε, είχε υποχρέωση βίζας, για τη Σερβία προχωρούμε προς ε, απελευθέρωση. Για δύο από τις τρεις λοιπόν ναι μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα, αλλά η τρίτη εθνότητα δεν θα μπορεί. Δύσκολο, δύσκολο να το υποστηρίξουμε. Πολλά από την έκθεση δεν θα μπορούσα να αλλάξω μάλλον, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε και να εκφράσουμε απόλυτα σαφώς τις θέσεις μας. Και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σαφείς στις θέσεις που εκφράζουμε. Δεν έχει νόημα να χαϊδεύουμε κανένα στα αυτιά, δεν έχει νόημα να είμαστε διακριτικοί και ευγενικοί. Νόημα έχει να στηρίξουμε το λαό, γιατί ο λαό έχει εμπιστοσύνη πιο πολύ σε εμά παρά στου ίδιου του πολιτικού, αν θέλετε να ξέρετε. Και γι' αυτό έχω και κάποιε προτάσει με τροπολογία, στην οποία απευθύνω έκκληση στο λαό να πάει στην κάλπη να ψηφίσει γιατί τους λέω εάν δεν πάτε στην κάλπη αφήνετε τη μοίρα σας στα χέρια εκείνων που μόνο με προπαγανδιστικό και λαϊκιστικό τρόπο προσπαθούν να επιβάλλουν τις δικές τους προτιμήσεις. Αυτό λέω προς όλο το λαό της Βοσνίας να είναι όλοι παρόντες στην κάλπη, να μιλήσει η λαϊκή βούληση και σε τελευταία ελάχιστα προκύψει και ένα πολύχρωμο αποτέλεσμα στις εκλογές, έτσι ώστε να εκφραστούν όλες οι τάξεις και οι θέσεις και οι εθνοτικές ομάδες ε, και όχι μόνο μία. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο κύριος Βόμποντα ήθελε κάτι να σχολιάσει. Να ψηφίσουν τους σωστούς, τους σωστούς υποψηφίους να ψηφίσουν. Μα σχεδόν οι πάντες είναι οι σωστοί ο πρόεδρος. Επόμενο θέμα πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία ένταξη του κόσμου πεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την ε, συνάδελφο Ουλρίκε Λούνατσεκ εντάχθηκε στην συζήτηση που έγινε για τα Βαλκάνια και στη συνέχεια η εισηγήτρια εισήγαγε ορισμένες τροπολογίες. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Λούνατσεκ, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ε, απόψε το απόγευμα θα συναντηθούμε με τον κύριο Σκέντερ Γιζενή, Υπουργό Εξωτερικών του Κωσυφοπεδίου. Δίνω το λόγο στην κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω αυτό το ημίωρο να έχουμε χρόνο για να παρουσιάσω την έκθεση και να σας ε, ρωτήσω πού συμφωνείτε και πού διαφωνείτε και που νομίζετε ότι υπάρχει αμφιγνωμία. Προσπάθησα στην ε, έκθεση αυτή, όπως είπε ο πρόεδρος, συζητήθηκε μέσα στα πλαίσια της ομάδας εργασίας για τα Δυτικά Βαλκάνια. Καταρχήν συζητήθηκε εκεί και στόχος ήταν να δούμε ότι το 2010 είναι κρίσιμο ε, για το Γιούλεξ, για την κυβέρνηση, για τις σχέσεις με τη Σερβία γιατί δύο χρόνια μετά από την ανεξαρτησία είναι κρίσιμο για τους πολίτες του Κωσυφοπεδίου να νιώσουν ότι η ζωή συνεχίζεται και γίνεται επιτελείται πρόοδος και στην καθημερινή του ζωή, διότι η ανεξαρτησία καθεαυτή δεν επιλύει τα, τα προβλήματα καθεαυτά. Υπάρχουν ε, επιτόπια προβλήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν. Ας ε, αρχίσω με τα βασικά σημεία δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί έχετε διαβάσει το κείμενο. Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημασία η ολοκλήρωση με τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η απελευθέρωση απελευθέρωση, η διαδικασία απελευθέρωσης ισχύει και για το κόσυφο πεδίο. Πιστεύω λοιπόν ότι από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιέσαμε εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή όλοι οι κάτοικοι της πρώην Λυκοσλαβίας να μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα με την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων και θα πρέπει να αρχίσουμε με τον οδικό χάρτη προς αυτή την κατεύθυνση μία μεγάλη μου ανησυχία, ένα μεγάλο μου μέλημα, γιατί βρέθηκα στο Κωσυφοπέδιο για τέσσερις μέρες την προηγούμενη εβδομάδα, στην τρίτη μου επίσκεψη σε αυτή τη χώρα, και αυτό δεν το ενέταξα στην ε, έκθεση, αλλά θα ήθελα να το πω, είναι το εξής. Δεν θα ήθελα να υπάρχει μία κοινή προσέγγιση με όλα τα κράτη-μέλη. Δεν πρέπει να αποδυναμώσουμε δηλαδή την υποστήριξη, δεν πρόκειται για Αλβανούς είτε για άλλες εθνότητες, θα πρέπει να την χάνουν τις ε, πλήρους υποστήριξής μας. Άρα θα πρέπει να έχουμε κοινή προσέγγιση για το κασοποπεδίο. διαφορετικά. Χάνουμε χρόνο, ε, χάνουμε χρήμα στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας. Αυτό όλο ένα και δυσχεραίνεται. Ενέταξα και τις σχέσεις μας με τη Σερβία. Ελπίζω να, έχουν, να υπάρξουν σχέσεις καλής γειτονίας στο μέλλον και ότι η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου ε, ε, είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Υπάρχουν και επικρίσεις ως προς τη, τη ε, διαφορετική αντιμετώπιση του καθεστώτος θεωρήσεων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, μερικοί ζητούν 60 ευρώ, να καταβληθούν 60 ευρώ και όχι 35, όπως ίσχυε, ε, θα έπρεπε να ισχύει για όλους. Μετά από τις πρώτες εκλογές πέρσι, τις δημοτικές εκλογές, οι οποίες δεν ενεργήθηκαν πολύ καλά, αυτό αναφέρεται στην έκθεση, θα ήθελα να προσθέσω και μία άλλη τροπολογία σε σχέση με την υποστήριξη της ε, ε, εκλεγμένης πλειοψηφίας του σερβικούς θύλακες. Υπάρχουν ε, παράλληλες υποδομές που υπάρχουν και ίσως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι προσδίδουμε μεγαλύτερη σημασία στο βορρά και όχι στο Νότο. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαία λοιπόν υποστήριξη παντού και η στρατηγική προς το είναι μια διαδικασία που έχει εκκινήσει και θα προσθέσω και μια άλλη τροπολογία για την ε, πίεση και εκφοβισμό στο, στο βόρειο τμήμα, δηλαδή οι Σέρβοι, οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν με τις αρχές του πεδίου. Αυτή δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Ως προς την επιτυχία του Γιούλεξ, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση, το προανέφερα και θα το αναφέρω και στον Υπουργό το απόγευμα. Η Γιούλεξ μπήκε και στο τομέα των μεταφορών και έγιναν έρευνες και στην οικία του Υπουργού Μεταφορών διότι ε, αναφέρθηκε ότι δυστυχώς έχει εμπλακεί σε περιπτώσεις διαφθοράς. Ελπίζω να ακολουθήσει την κανονική δικαστική οδό αυτή η διαδικασία με βάση τις προσταγές της Γενικής Εισαγγελίας. Η υπόθεση Άλβιν Κούρτε αναφέρθηκε ως προς την πολιτικοποίηση της υπόθεσης αυτής. Μίλησα για τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης. Αυτό το ανέφερε και η Doris Πακ, καθώς και το θέμα της ε, εκπαίδευσης και το γλωσσικό ε, ζήτημα και σύστημα και τα προβλήματα μεταφοράς και ενέργειας. Θα πρέπει να αναφερθούν εδώ. Θα σταματήσω εδώ για να ακούσω τα δικά σας σχόλια και να μην σας διαβάζω τμήματα της έκθεσης. Ευχαριστούμε. Πανσέρι ε, από τους κοιόδης των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ορισμένες ε, σκέψεις μόνο, γιατί η κυρία Λούνατσεκ επετέλεσε μια πολύ καλή εργασία και νομίζω μπορούμε να δεχτούμε τα περισσότερα σημεία έτσι ώστε να γίνουν βήματα προς τα εμπρός και το κοσυβοπαίδιο να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη χώρα αυτή σε στάση αναμονής, διότι αυτό θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στο, στην υπόλοιπη ε, περιφέρεια των Δυτικών Βαλκανίων. Άρα δεν μπορούμε να προωθήσουμε μία ε, σχηνοτενή συζήτηση και θα πρέπει να προωθήσουμε τη σταθερότητα στην περιφέρεια αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ο βασικός παράγων δράσης υπέρ αυτής της πορείας. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια ιδεώδη κατάσταση, όμως δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική παρά να ενταχθεί το κοσυφοπέδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τουλάχιστον εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υπάρχει μια κοινοτική θεώρηση και όχι διακυβερνητική. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να επιλύσουμε θέματα που άπτονται της ε, χρηματοπιστωτικής ε, κρίσης και σε αυτές τις χώρες. Τώρα, ως προς τις προσεγγίσεις της κυρίας ε, Λούνατσεκ, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν ορισμένα σημεία όπου θα πρέπει να δοθούν ορισμένες διευκρινήσεις για να ανταποκριθούμε στους στόχους, στους αρχικούς στόχους. Το πρώτο σημείο αφορά το σημείο που καλούμε τα κράτη-μέλη, ε, ακόμα και αυτά που δεν έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του κόσυφο πεδίου, να προωθήσουν μία κοινή προσέγγιση. Κοινή προσέγγιση γιατί όμως. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να εντάξουμε το γεγονός ότι αυτή η κοινή προσέγγιση θα πρέπει να ξεκινά από τη σκέψη ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο μη επιστροφής. Διαφορετικά ποια θα είναι η κοινή προσέγγιση. Ένα δεύτερο θέμα αφορά την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας ένταξης, στα πλαίσια και των σχέσεων καλής γειτονίας. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ εξέλιξης του κοσυφοπεδίου και υποψηφιότητας της Σερβίας προς για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί θεωρούν ότι δεν υπάρχει συσχετισμός, εγώ όμως τον υποστηρίζω. Αυτή τη συνάφεια δηλαδή. Επίσης, εφήγει το θέμα και πολύ σωστά ορισμένων ανησυχιών ως προς τη δράση της Ιούλεξ σε σχέση με τους στόχους που είχαμε θέσει για τη δράση της Ιούλεξ. Δεν ξέρω κατά πόσο η διατύπωση είναι ευτυχής, αλλά θα ήθελα να προτείνω τη σύσταση μιας επιτροπής ad hoc με εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κομισιόν για να δούμε πώς προωθούνται οι δραστηριότητες της Γιούλεξ, διότι από αυτό εξαρτάται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την περιοχή. Και θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι η εργασία της κυρίας Λούνατσεκ ήταν εξαιρετική. Ωραία. Έχουμε τις άλλες παρεμβάσεις τώρα για δύο λεπτά ο καθένας. Ο κύριος Ντανζάν έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ. Καταρχήν συγχαρητήρια κυρία Λουνατσέκ. Καταπληκτική και πολύ αξιόλογη έκθεσή σας για μια πολύ περίπλοκη και λεπτή κατάσταση. Δύο ίσονο σημασίες θέματα καταρχήν και μετά δύο πιο σημαντικά. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι χάρη στην Καφόρ, χάρη στη Γιούλεξ και στην κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου, αλλά και χάρη στην ε, κυβέρνηση του Βελιγραδίου, που δεν ε, κατέφυγε σε προβοκάτσιες, αλλά χρησιμοποίησε μόνο τη διπλωματική οδό για τα θέματα τη ε, ανεξαρτησία. Όλα αυτά διασφάλισαν την σταθερότητα στο Κωσυφοπαίδιο, παρόλο που πολλοί, ιδιαίτερα από τι χώρε που δεν αναγνώρισαν την ανεξαρτησία, προέβλεψαν ε, χάο και δυσλειτουργιακά που αποφεύθηκε. Για την περίπτωση Κούρτη θα ήθελα να πω το... ότι είναι υπερβολική αυτή η αναφορά, γιατί έτσι κάνουμε τη διαφήμιση σε κάποιον που δεν αξίζει τέτοια απήχηση και προβολή πραγματικά. Ας μην κατονομάσουμε την υπόθεση Κούρτη. Πολύ σημαντικό το σημείο 4 για τις σχέσεις με τη Σερβία. Νομίζω ότι είναι καθήκον μας να δούμε και το μέλλον. Όπως είπατε, δυστυχώς είναι ανύπαρκτες οι σχέσεις με τη Σερβία. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε το διάλογο μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Σερβίας. Γνωρίζουμε όλοι ότι θα είναι περίπλοκος ο διάλογος σε πολιτικό επίπεδο, αλλά τουλάχιστον να ενθαρρύνουμε το διάλογο σε λειτουργικό επίπεδο και κατόπιν θα φτάσουμε ίσως σε πολιτικό διάλογο. Θα, θα πρέπει και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαιτήσει αυτό το διάλογο, γιατί είναι αδιανόητο παρά τις δυσκολίε να μην μιλούν αυτοί οι δύο λαοί μεταξύ τους. Άλλωστε οι θύνοντες του Κωσυφοπεδίου είναι οι πολύ ανά πάση στιγμή μπορούν να γίνουν το αντικείμενο ενταλμάτων σύλληψης. Δεν νομίζω ότι είναι ε, καλή αυτή, καλός αυτός ο χειρισμός ε, για αγαστές διπλωματικές ε, σχέσεις. Και δεν νομίζω ότι είναι δόκιμο να επαπειλείται έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά εθνών των για αποσχιστικές απόπειρες κτλ. Η κατάσταση στο Βορρά είναι πολύ ιδιάζουσα και πολύ ευαίσθητη η απόσχηση του βόρειου τμήματος δεν είναι αναλλακτική λύση και πολλοί ε, στο Βελιγράδι δελεάζονται από αυτή την πιθανότητα. Επίσης είναι σωστή μια σταδιακή προσέγγιση για το Βορρά. Αυτοί που ζητούν ε, μαζική παρουσία ε, της διεθνούς κοινότητας στο Βορρά προκειμένου να επανέλθει το συντομότερο δυνατό δεν είναι σωστή προσέγγιση. Το σχέδιο της Άρη ήταν πολύ καλό από πολλές απόψεις και είχε πολύ σωστούς μηχανισμούς. Νομίζω ότι είναι βάση για έναν επιχειρησιακό, λειτουργικό διάλογο μεταξύ Πριστίνα και Βελιγραδίου. Κύριο Σεβερή, τρεις παρατηρήσεις κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν πιστεύω ότι πριν να μιλήσουμε για την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση του Βοσυφοπεδίου, καλό θα ήταν να μιλήσουμε για την συνδρομή προς το κοσυφοπαίδιο, ώστε να μετατραπεί σε μια σύγχρονη οντότητα αυτοσυντηρούμενη. Αυτή είναι η πρώτη επιτακτική ανάγκη και μετά να, ζητήσουμε, να μιλήσουμε για την εσωμάτωση του κοσυφοπαιδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι υπάρχει μια σύνδεση, μια διασύνδεση μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου όταν μιλούμε για θέματα ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης και ευρωπαϊκών σχέσεων. Αυτή η διασύνδεση όμως, αυτή η σχέση δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να θέσουμε όρους στη Σερβία ανάλογα με την πολιτική της προς το Κωσυφοπέδιο και αυτή η πολιτική να γίνει όρος για την ε, ένταξη της Σερβίας. Δεν είναι αυτή η σωστή διασύνδεση. Το ζητούμενο είναι να βρούμε μια λύση για ολόκληρη την περιοχή προκειμένου να επανέλθει το σύνολο της περιοχής στο δρόμο της διεθνούς νομιμότητας, κάτι που δεν έχει επιτευχθεί ακόμη, και μιας ε, πολιτικός ε, ορθολογικής λύσης. Και το τρίτο μου σχόλιο είναι ότι θα πρέπει να αποφύγουμε την πολιτική της τρουθοκαμήλου που δυστυχώς ε, αντανακλάται στην έκθεση κατά κάποιο τρόπο. Το πρόβλημα μα είναι ότι δεν έχουμε κοινή θέση για το κοσυφοπαίδιο και δεν μπορούμε να ζητήσουμε από αυτού που αναγνώρισαν την ανεξαρτησία του κοσυφοπαιδίου να την αποσύρουν ή να ζητήσουμε από αυτού που δεν αναγνώρισαν το κοσυφοπαίδιο να το αναγνωρίσουν για να βρούμε λύση. Ούτε το status είναι λύση, ούτε η παρούσα κατάσταση είναι λύση. Και για να έχουμε μια κοινή προσέγγιση, όπω είπε σωστά ο κ. Παντσέρη, θα πρέπει να έχουμε και ένα κοινό πρόγραμμα για το μέλλον. Για το μέλλον όμω, όχι για το παρελθόν. Και από αυτή την άποψη θα ήθελα στην έκθεση να προδιαγράφονται διάφορες ε, ιδέες για να μας δίνουν μια γενική κατεύθυνση. Ποιος είναι ο απότερος σκοπός μας. Δεν μπορούμε να βρούμε λύση κατατεμαχισμένη, αποσπασματική, αναζώνη, αναπεριοχή. Χρειαζόμαστε μια περιφερειακή προσέγγιση και ένα πακέτο, μια συνολική λύση. Το λόγο ο κύριος Μούνιτς. Κυρία, συγγνώμη, Μουνίθ. Ε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριο Σέβερεν. Η σταθερότητα στην περιοχή και μια φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση στο, στη Σερβία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό ότι πολλέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλέ χώρε τη παγκόσμια κοινότητα δεν αναγνώρισαν το κοσυφοπαίδιο την ε, μονομερή ανακήρυξη ανεξαρτησίας χωρίς συμφωνία μεταξύ των μερών και χωρίς ε, απόφαση, μάλλον ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Γιατί λοιπόν οι χώρες ε, να αναγνωρίσουν το κοσυφοπαίδιο δεν εκπληρώθηκαν αυτές οι δύο προϋποθέσεις. Ούτε μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητά από τις χώρες που δεν αναγνώρισαν το κοσυφοπαίδιο να το κάνουν. Άλλωστε, ακόμη και μια αναγνώριση ε, προ, δίνει μια προστιθέμενη αξία, φέρνει την ε, κυβέρνηση της Σερβίας πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτή την άποψη, ο τρόπος που αναφερόμαστε στο κοσυφοπαίδιο σε όλες τις σχετικές εκθέσεις θα πρέπει να είναι ε, ο, ο τρόπος που υιοθετούμε στις άλλες εκθέσεις, όπως το ταζόν και Φεζόν, για την, για την απελευθέρωση του κοσυφοπεδίου. Να αναφέρουμε το πώς αναφέρεται το κοσυφοπαίδιο στο ψήφισμα 1244 του ΟΗΕ. Αυτή να είναι η ονομασία που θα χρησιμοποιούμε σε όλες μας τις εκθέσεις. Αυτή που αναφέρεται στο ψήφισμα ασφαλείας 1244 του ΟΗΕ. Ευχαριστώ την κυρία Λούνατσεκ. Ήταν επικοδομητική η θέση της γενικώ, αλλά προσοχή, θα πρέπει να προσέξουμε ορισμένα θέματα του κοσυφοπεδίου και της ε, διεθνούς νομιμότητα. και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ζητούμε από τι χώρε μέλη να αναγνωρίσουν ε, τη χώρα αυτή εφόσον δεν πληρούνται οι προποθέσει ε, του ΟΗΕ. Ο κύριος Κατσίν, αλλά πρώτα θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα το απόγευμα θα αρχίσουμε στις 3 και 4 και όχι στις 3 ακριβώς. 3 και 4 λοιπόν με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κωσυφοπεδίου. 3 και 4 ραντεβού το απόγευμα και όχι 3 ακριβώς. Και πρώτο θέμα θα είναι η συνάντηση με τον υπέξ του Κωσυφοπεδίου. Ο κύριος Κάτσιν. Σας ευχαριστώ. Η ανάγκη διαλόγου μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Σερβίας είναι προφανής, αλλά θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Ντανζάν, που είπε ότι είναι δύσκολο να προωθήσουμε σχέσεις μεταξύ γειτονικών χωρών αν δεν υπάρχει διάλογος. Είναι δύσκολο όμως να ε, υπάρχουν ε, γειτονικές σχέσεις εφόσον η Σερβία χαρακτηρίζει το κοσυφοπαίδιο όχι γειτονική χώρα αλλά τμήμα της. Είναι ασαφή τα πράγματα και η κατάσταση. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι, πώς θα ξεκαθαριστεί η κατάσταση και ευελπιστώ ο διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας να οδηγεί σε συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων των δύο χωρών στη συνδιάσκεψη του Σεράγεβο της Δευτέρας Ιουνίου. Είναι σημαντικό θέμα ο διάλογος για να επιτευχθεί πρόοδος. Επίσης υπάρχει το δίλημα της συμμετοχής αφενός και της απομάκρυνσης αφετέρου ή της περιθωριοποίησης. Οι Σέρβοι έχουν τη δική τους τοπική διοίκηση, η οποία δεν έχει καθόλου πόρους. Και τώρα που ανέλαβαν την εξουσία θα μπορέσουν να κάνουν αυτά που περιμένει ο λαός. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την χρηματοδότηση της σερβικής κοινότητας στο Κωσυφοπαίδιο, ώστε

Το θέμα της ε, απελευθέρωσης των ε, θεωρήσεων είναι θέμα τήρησης υποσχέσεων, γιατί και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσαν σχετική υπόσχεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γι' αυτό και θα πρέπει να απαιτήσουμε από τα δύο θεσμικά όργανα να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Συγχαρητήρια κυρία Λούνατζε και ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας. Το λόγο κύριο Στάλερ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Λούνατσεκ, την εισηγήτρια, διότι αντιμετώπισε αυτό το, το θέμα παγίδα κατά πολύ καλό τρόπο το κοσυφοπέδιο βαραίνει πολλές χώρες ε, και αυτό μπορώ να το πω χωρίς καμία αμφιβολία. Αυτό ίσχυε ε, ήδη από την εποχή της ε, Ιουκοσλαβίας η Σερβία του Μιλόσεβιτς στην ουσία απομάκρυνε τους ε, Αλβανούς βία. Γι' αυτό τώρα έχουμε έναν εξάρτητο κοσυφοπέδιο και θα πρέπει να αρχίσει να μας απασχολεί το θέμα από αυτή την οπτική γωνία και θεώρηση η Πρίστινα και το Βελιγράδι θα πρέπει να ξεκινήσουν έναν διάλογο και η καλύτερη προσέγγιση είναι να είμαστε πραγματιστές. Δεν υπάρχει άλλη λύση δυστυχώς έμπρακτα το κοσυφοπέδιο και η Σερβία θα επανενωθούν κατά κάποιο τρόπο όταν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι το ερώτημα ρητορικό να ρωτάμε τι θα συμβεί αν το Κωσυφοπέδιο ξαναενταχθεί στη Σερβία. Και θα ήθελα να συγχαρώ τους ιτήνοντες στο Βελιγράδι, διότι ε, ήταν ιδιαίτερα ορθολογική. Όμως αυτός ο διάλογος πρέπει να προωθηθεί. Θα πρέπει να ασχοληθούν με πρακτικά ζητήματα. Θα ήθελα να ευχηθώ στην Ισπανική Προεδρία κάθε επιτυχία για την διενέργεια της διάσκεψης στο Σαράγεβο. Ήταν μεγάλο λάθος που δεν λάβαμε υπόψη τη διάσκεψη στη Σλοβενία, στο Μπρντό, στο τέλος του, του μήνα. Τώρα όμως η Προεδρία που δεν επιτέλεσε το έργο της αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή πώς να βρεθούν σε κοινό έδαφος η Πρίστινα και το Βελιγράδι και ελπίζω να βρεθεί μια σωστή κοινή, αποδεκτή λύση. Η κυρία Κοπά. Ε, Νικολάη και Τόκες. Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Λούνατσεκ για την ειλικρινή της προσπάθεια να διαχειριστεί ένα τόσο σύνθετο ζήτημα και όπως είπε ο συνάδελφος Στάλλερ είναι πραγματικά μια καυτή πατάτα για το Ευρωκοινοβούλιο στο οποίο όλοι γνωρίζουμε τις συζητήσεις που είχαν γίνει όλα και τις συγκρούσεις τα περισσότερα χρόνια για το θέμα του καθεστώτος. Το βασικό σε μια έκθεση του Κοινοβουλίου για το Κόσοβο πρέπει αυτή τη στιγμή να είναι να τονιστούν οι κοινοί τόποι όπου μπορούμε να συναντηθούμε όλοι. Και αυτοί που έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσόβου και αυτοί οι οποίοι δεν την έχουν ε, αναγνωρίσει. Γιατί ε, νιώθω υποχρεωμένη να επαναλάβω για άλλη μία φορά ότι οι χώρες δεν γίνονται ανεξάρτητες με πλειοψηφίες, αλλά σύμφωνα με κανόνες του διεθνούς δικαίου, που ακόμα δεν, τους, δεν συναντιούνται οι όροι αυτοί στην περίπτωση του Κωσόβου. Έτσι λοιπόν το θέμα της νομικής βάσης, την οποία περιλαμβάνει η κυρία Λούνατσεκ στο κείμενό της, είναι πάρα πολύ βασικό. Και θα συμφωνήσω με την άποψη της ε, συναδέλφου Νίζου, ότι πρέπει να αναφέρεται το Κόσοβο σύμφωνα με το 1244. Από εκεί και πέρα. Είναι πραγματικά μεγάλος ο προβληματισμός όταν εξετάζουμε το θέμα του Κόσοβου και της Σερβίας. Ε, η Σερβία, όπως όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ήταν υποχρεωμένη να δεχθεί έναν επιπλέον όρο, ένα επιπλέον κριτήριο ένταξης, που ήταν ε, η συνεργασία με το δικαστήριο, ποινικό δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία. Τώρα βλέπουμε de facto να δημιουργείται ένας νέος όρος που είναι η αναγνώριση του Κωσόβου. Πρέπει να προσέξουμε να μην αυξήσουμε τις πιέσεις στην πιο ευρωπαϊκή κυβέρνηση που είχε ποτέ η Σερβία, ώστε να ξεπεραστούν τα όρια που εκείνη μπορεί να αντέξει. Το θέμα της Γιούλεξ. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον συνάδελφο Ντανζάν ότι πρέπει να επιμείνουμε στη σταδιακή ε, εφαρμογή του προγράμματος της Γιούλεξ. Αλλιώς οι αντιδράσεις θα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλες. Νομίζω η προσοχή και η ευαισθησία στα τοπικά θέματα με την οποία έχει κινηθεί μέχρι τώρα η Γιούλεξ έχει εμποδίσει να ε, έχουμε επανάληψη συγκρούσεων και νομίζω ότι αυτό είναι ο δρόμος στον οποίο πρέπει να πορευτούμε. Τέταρτο σημείο, οργανωμένο έγκλημα. Ε, στο άρθρο 9 βλέπουμε ότι υπάρχει μία αναφορά στο οργανωμένο έγκλημα μόνο στο βορρά της περιοχής. Θα ήθελα μία απάντηση για την κυρία Λούνατσα, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το οργανωμένο έγκλημα αφορά όλο το Κόσοβο και όχι μόνο το Βορρά. Και τέλος, θέμα πολιτιστική κληρονομιάς. Θα ήθελα να υπάρχει στο κείμενο μία παράγραφος για την ανάγκη αποτελεσματική προστασία της πολιτιστική κληρονομιά στο Κόσοβο, με ιδιαίτερη προσοχή για τα σερβικά ορθόδοξα μοναστήρια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να είσαστε ιδιαίτερα Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα επιχειρήσω μια πολιτική προσέγγιση γιατί ίσως υπερπολιτικοποιήσουμε τα πράγματα. Θα επικεντρωθώ και θα περιοριστώ στους κανόνες διεθνούς και κοινοτικού δικαίου. Είναι αμφισβητήσιμο το νομικό καθεστώς του κοσυφοπεδίου με βάση τους διεθνείς κανόνες και μάλιστα αναμένεται νομική γνωμοδότηση, την περιμένω. Τότε θα δούμε σε ποιο βαθμό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διεθνείς κανόνες για την κοινότητα. Και μπορούμε να μιλούμε για το θέμα μόνο εφόσον δεν ε, ε, καταστρατηγήσουμε τα κριτήρια της Κοπενχάγης που θα πρέπει οπωσδήποτε να εκπληρώνονται για να είναι επιλέξιμο ένα κράτος για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Δεν είναι απόλυτα ορθή η προσέγγιση της κυρίας Λούνας εξ' ό,τι αφορά την κατάσταση στο κοσυφοπαίδιο. Πάντως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι εξασφαλίζεται σε πολιτικό επίπεδο η σταθερότητα του κοσυφοπεδίου, αλλά η πολιτική σταθερότητα είναι επισφαλής ακόμη και για χώρες που είναι ασφαλείς, ε, σταθερές από κοινωνική και κοινωνική άποψη. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτε για οικονομία της αγοράς, ούτε για γνήσια οικονομία στο κοσυφοπέδιο. Αλλά και στα κοινωνικά θέματα υπάρχει πρόβλημα. Η ανεργία καλπάζει και έχει φτάσει στο 40%. Και σίγουρα η σταθερότητα του κοσυφοπεδίου επηρεάζει τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Επίσης ε, υπάρχουν θέματα διακυβέρνησης και τα κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος που δρούν όχι μόνο στην περιοχή αυτή αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ίσως και εκεί δημιουργηθούν ερωτηματικά για το νομικό καθεστώς. Είμαστε υπέρ της σταθερότητας στην περιοχή, είμαστε υπέρ της συνεργασίας, αλλά σημαντικό για μας ε, είναι να τηρηθούν οι διεθνείς κανόνες. Αυτό μας ενδιαφέρει ως ε, Ευρωπαίους. Um, um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχει επιτελεστεί εξαιρετική εργασία από τη συνάδελφο Ουλρίκε, αλλά πέραν από, πέρα από την έκθεση αυτή, νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα της Σερβίας και του Κόσυφο πεδίου ως προς την ένταξή τους. Αυτά τα δύο ζητήματα δεν μπορούν να διαχωριστούν. διότι το κοσυφοπέδιο θα πρέπει να μας απασχολήσει υπό το φως ε, του κομμουνιστικού καθεστώτος που κάποτε διακυβέρνησε αυτή τη χώρα, διότι αυτό είναι κληροδότημα αυτής της κατάστασης του παρελθόντος. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι αυστηρότερα ως προς την ένταξη της Σερβίας, αλλά η Σερβία είναι το κλειδί για το κατά πόσο θα υπάρξει ειρήνη στο Κωσιβοπέδιο. διότι εάν η Σερβία δεν ενθαρρύνει του Σέρβους του Κωσυφοπεδίου να καταδείξουν μια συμφιλιωτική στάση, τότε δεν θα επιτύχουμε τίποτα. Μόνο αν υπάρξει μια πραγματική συμφιλίωση, μια βελτίωση της κατάστασης, θα φτάσουμε σε κάτι το χειροπιαστό. Εδώ δεν φτάνουμε σε συμφωνία μεταξύ των 27 κρατών μελών. Εγώ είμαι Ούγγρος από την Ρουμανία και η Ρουμανία δεν αναγνωρίζει το κοσυφοπέδιο. Άρα αν δεν φτάσουμε σε συμφωνία μέσα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για το κοσυφοπέδιο, τότε πώς να συμφωνήσουν αυτές οι δύο χώρες μεταξύ τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο με την Ισπανική Προεδρία για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση του κοσυφοπεδίου κυρίως από τη Σερβία. Και αυτό είναι το θέμα ουσίας. Πριν από τα συμπεράσματα της ε, εισηγήτριας της κυρίας Λούνατσεκ, Έχουμε τον κύριο Μιρέλ από, τον, ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ήθελα να είναι ιδιαίτερα σύντομος, δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστώ την κυρία Λούνατσεκ για την εξαιρετική έκθεση. Συμφωνούμε απολύτως το 2010 είναι το κλειδί για το κοσμοπέδιο. Όσο όμως για το κοσμοπέδιο είναι και για μας έτος κλειδί και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε πολλές πρόοδους. Η Πρίσνα θα πρέπει να προχωρήσει πολλές μεταρρυθμίσεις και ναι υπάρχει υποχρέωση, η δέσμευση για την απελευθέρωση της διαδικασίας για τη διαβατηρίου με προϋπόθεση όμως, ή προϋποθέσεις καλύτερα, την συμφωνία περί επανεισδοχής και της, ε, την εξασφάλιση των συνθήκων εκείνων που θα επέτρεπαν την ε, επανένταξη, την επανενσωμάτωση της κοινωνίας τους των επαναπατρισσομένων. Και εάν αυτό συμβεί, τότε με τον Ιούνιο θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία για την απελευθέρωση. Για το βορρά της χώρας και άνοιξε ο οίκος Ευρώπης και χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και 3-4 χρόνια ε, διάφορα σχέδια στην περιοχή, στο βορρά, δηλαδή έχουμε σαφή παρουσία εδώ και χρόνια. Και για να απαντήσω στον κύριο Κατσίν, πριν από λίγο διάστημα προσεφέρθηκε χρηματοδοτική υποστήριξη στους πρόσφατα εκλεγέντες δημοτικούς και τοπικούς εκπροσώπους για την υποστήριξη της του έργου τους. Ε, και κατά τα άλλα, ναι, έχουμε μέτρα χάρη στο έλεξ που μας επιτρέπουν να ολοκληρώσουμε έργο σημαντικό για τα τελωνία, για την αστυνομία, για την επανενσωμάτωση στο αστυνομικό σωματικό του των Σέρβων του Κοσμοπεδίου, το, την επανέναρξη του δικαστηρίου της Μητρόβιτσα, αλλά δεν είναι εύκολο βέβαια να ανοίξει φάκελος ε, για την καταπολέμηση διαφθορά, σε παραδείγματι. Δεν μπορεί, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με άλλες υποθέσεις, να πούμε ότι από τη μια μέρα στην άλλη προχωρούν ε, οι δικαστικές αυτές διαδικασίες, γιατί χρειάζονται και αποδείξεις και στοιχεία και τεκμήρια και όλα αυτά. Και Συμφωνώ με τον κύριο Τόνζον για να κλείσω ότι όλοι οι Κασάνδρες διαψεύστηκαν γιατί το κοσφοπέδιο επέζησε και προχωράει. Ε, για να κλείσουμε λοιπόν η κυρία Λούνατσικ. και σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ για τα σχόλια όλους τους συναδέλφους, για τις παρατηρήσεις, για τα αιτήματα που ακούστηκαν. Πολύ ευχαρίστως θα τα λάβω υπόψη ή τουλάχιστον θα τα συζητήσω μαζί γιατί σε ορισμένα δεν θα συμφωνήσω όπως θα φαντάζεστε ενδεχομένω, με άλλα όμως θα συμφωνήσω. Και θα συνομιλήσω με όλους τους κοιοδησιτές πριν από το ΙΝ προθεσμία 18 Μαΐου για την κατάσταση των τροπολογιών για να λύσουμε το πρόβλημα και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρεται παρακαλώ να μου ε, μιλήσει εφόσον θεωρεί κάτι σημαντικό. Ήταν πολύ σημαντική η εμπειρία αυτή για μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αλλά και τη, όλους σας, αλλά και την Εύα Μάρ και το προσωπικό μου όλο που με βοήθησε ιδιαίτερος ε, στην προσπάθεια αυτή. Για τώρα, για το περιεχόμενο. Σε ένα βαθμό θα αναφερθώ μόνο, ο κ. Ντανζάν αναφέρθηκε στην ανάγκη διαλόγου μεταξύ ε, Κοσφοπεδίου και Σερβίας. Συμφωνώ σε αυτό, το θέμα είναι ποιος θα συνομιλήσει με ποιον. Ιδιαίτερα σημαντικό βρίσκω το να υποστηριχθεί ο διάλογος σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών και από εκεί να πιεσθούν και οι κυβερνήσεις. Και βέβαια πρέπει να ενισχυθεί και η ευρωπαϊκή πλευρά. Σε σχέση με τη δικαστική υπόθεση που ακούστηκε νωρίτερα, να έχω συζητήσει πολύ με αρκετούς, ωστόσο το κενό που η προσφορά μάλλον βοήθησε από την Έλεξ τον στήριξε αρκετά τον κύριο αυτόν και έτσι πιστεύω ότι θα υπάρξει δυνατότητα και για άλλους να μπορέσουν ε, να να επωφεληθούν τις ίδιες υποστήριξη. Υπάρχει πολλή πολιτικοποίηση γύρω από την υπόθεση αυτή. Επίσης υπόθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξουν, να επιβληθούν επιπλέον όροι στη Σερβία σε σχέση με την αναγνώριση του Κοσμοποδίου. Θα πρέπει να πω ότι και εγώ ήμουν μάλλον επικριτική ως προς τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια αυτή η διαδικασία. Τώρα όμως νομίζω ότι πρέπει να πιέσουμε τη Σερβία. Δεν θέλουμε κι άλλη Κύπρο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα συμφωνήσω λοιπόν με αυτή την τοποθέτηση. Γιατί κάνει κακό σε όλες μας προσπάθειες, ε, ζημιώνει κάθε μας προσπάθεια εκεί και ναι, δεν είναι αναγκαίο να πιέζουμε τόσο πολύ πάντοτε, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι ένας όρος και για την Ευρωπαϊκή Ένωση τελευταία ανάλυση και λυπούμε αν είμαι τόσο πια ομή. Κάποιο άλλο μίλησε για πολιτική στρουφοκαμήλου στην έκθεση. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω διότι τελικά δεν ζητάω τρει διευθύνσει ούτε ζητώ από τους, 5, ε, από τους 22 να ανακαλέσουν την ε, ε, αναγνώριση του Κοσμοπαιδίου, ούτε απαιτώ από τους 5 που δεν έχουν αναγνωρίσει να το αναγνωρίσουν. Θα ήθελα φυσικά, αλλά δεν μπορώ να τους υποχρεώσω. Επίσης, ο κύριος Τάλερο, ο κύριος Κάτινερ αναφέρθηκαν στην διάσκεψη για το Σαράγεβο. Ναι, δεν έχει όμως θέση μέσα στην έκθεση. Παρ' όλα αυτά ελπίζω να στεφθεί με επιτυχία. Ελπίζω η Ισπανική Προεδρία να μπορέσει να φέρει καλά αποτελέσματα. Για το Γιούλεξ νομίζω που μίλησαν όλοι. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε εδώ σύγκρουση, διαφορά με τους, ε, με Αμερικανούς και θα πρέπει να δούμε πώς θα υποστηριχθεί η Γιούλεξ. Ο κύριος Μιρέλ μίλησε για τη διαδικασία απελευθέρωση των ε, ε, θεωρήσεων διαβατηρίων. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μιρέλ για την υπόσχεση της δεσμεύσης και ελπίζω ότι θα ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι ναι, Βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα. Όλοι οι υπουργοί με του οποίου όμω έχω συνομιλήσει στο Κοσμοπέδιο δηλώνουν την ίδια βούληση. Λένε θέλουμε να προχωρήσουμε, θέλουμε να το υπογράψουμε, θέλουμε να μπορούμε να ε, υλοποιήσουμε τη συμφωνία επανεισδοχή. Όμω δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα. Δεν έχει το κόσμο αρκετά χρήματα. Προσπαθούν και ιδιαίτερα για του Ρωμά. Κάνουν ιδιαίτερε προσπάθειε, αλλά δεν ε, υπάρχουν τα χρήματα. Και εδώ επικρίνω εγώ τα κρατημέλη, γιατί δεν βλέπω γιατί 10.000 εκτοπιστέντε στη Γερμανία μπορεί να είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα για μια χώρα τόσο μεγάλη. Ενώ εάν πάνε χωρίς ε, τους κατάλληλους όρου στο κοσφοπέδιο, προφανώς θα σημαίνουν σημαντικές ε, δυσκολίες. Αλλά πάντως, όπως είπα, ελπίζω να ικανοποιηθούν όλοι οι όροι ώστε να ξεκινήσει μαζί με το φιλοπορία η διαδικασία.